Okay, colleagues, can we, can we begin? Firstly, let me give uh apologies. Ο Μπέρν ζητά συγγνώμη γιατί κολλείεται σήμερα. Οπότε εγώ ως πρεσβύτερος θα προεδρεύσω γιατί ούτε οι αντιπρόεδροι είναι ελεύθεροι σήμερα. Σε ό,τι αφορά την έγκριση της ημερήσιας διάταξης, έχω δύο προτάσεις. Οι πράσινοι ζήτησαν αναβολή του σημείου 16. Προτείνω να συμφωνήσουμε για την αναβολή του 16. Οι μεταρρυθμιστές και συντηρητικοί ζήτησαν αναβολή των ψηφοφοριών. Αυτό το έτοιμο είναι πιο προβληματικό. Γιατί από τις 28 Οκτωβρίου υπήρχε η ημερήσια διάταξη και μόνο χθε υπευλήθη το, το αίτημα αναβολής και ιδιαίτερα αν δεν ψηφίσουμε για την πολιτική ανταγωνισμού, θα χάσουμε την ευκαιρία να επιδώσουμε εγκαίρως τη γνωμοδότησή μας. Οπότε εγώ είμαι κατά της αναβολής, αλλά με βάση τον κανονισμό πρέπει να ψηφίσουμε προ προς το αίτημα της ECR. Ερωτώ λοιπόν, είναι κανείς υπέρ της αναβολής των ψηφοφοριών. Κατά της αναβολής αποχές είναι σαφές ότι απορρίπτεται το αίτημα των ECR, άρα θα ψηφίσουμε σήμερα. Υπάρχουν άλλα σχόλια για την ημερήσια διάταξη. Αν όχι, θεωρώ ότι εγκρίνεται. Πρακτικά, της 15ης Οκτωβρίου. Τα έχετε λάβει, οπότε αν δεν υπάρχουν σχόλια μέχρι το τέλος της συνεδρίασης, θα θεωρηθούν συγκεκριμένα. Σημείο 3, ανακοινώσεις του Προέδρου. συνήθεις ανακοινώσεις, δηλαδή αναμεταδίδεται από το διαδίκτυο η συνεδρίαση οπότε και οι διερμηνείς σας παρακαλούν να μιλάτε με κανονικό ρυθμό γιατί συνήθως ε, μιλάτε με μεγάλη ταχύτητα. Αγαπητέ Πρόεδρε, ένα σημείο θα ήθελα να δείξω για σήμερα αν θα μπορούσαμε σε μία από τις επόμενες συναντήσεις των συντονιστών να το συντήσουμε και με τον Πρόεδρο. Έγινε μία διάσκεψη αυτή την εβδομάδα όπου πήρε το λόγο και ο Πρόεδρος για την ε, ΣΥΤΑ και για την προστασία των επενδυτών. Στην ομάδα μας υπάρχουν διάφοροι συναδελφοί που έχουν την εντύπωση ότι ο Πρόεδρος δεν εκφράζει απαραίτητα την πλειοψηφία ε, της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου, αλλά πιο πολύ την άποψη της ομάδας τους και θα θέλαμε να συζητήσουμε για να δούμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τέτοιες περιπτώσεις και περιστάσεις. Αν θα μπορούσαμε να το θέσουμε λοιπόν το θέμα σε κάποιες ε, από τις επόμενες συναντήσεις, συνεδριάσεις, επειδή αυτό το θέμα προβλήθηκε και στον τύπο, ότι υπάρχει διαφορά απόψεων σε πολλά ζητήματα. Ο Πρόεδρος θα το αποφασίσει. Ε, μετά από τη συζήτηση στη συνεδρίαση των συντονιστών. Μία ανακοίνωση έχω μόνο ε, για την εξαίρεση σε ό,τι αφορά τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες. Χθε ανακοινώσαμε στον ΠΟΕ ε, τις προ, προτιμησιακές ρυθμίσεις ε, για τις υπηρεσίες σε ό,τι αφορά τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες. Η εξαίρεση αυτή είναι πολύ σημαντική και αναφέρθηκε και στην Διευπουργική του Μπαλή. Και η εξαίρεση θα διαρκέσει μέχρι ότου μια χώρα εξέλθει από την ομάδα των χωρών των λιγότερων ανεπτυγμένων, των ΛΑΧ. Σε ό,τι αφορά τι διαπραγματεύσει τριμερούς διαλόγου δεν είχαμε από την προηγούμενη συνεδρίαση τριμερή διάλογο, οπότε δεν έχουμε θέμα ενημέρωση. και περνάμε στα κυρίω θέματα την κοινή συζήτηση για τα σημεία 5 και 6, τη ρήτερης διασφάλισης και μηχανισμό κατά της στρατη... για τη Μολδαβία και τη Γεωργία. Σε ό,τι αφορά τις προτιμής συμφωνίας συμφωνία σύνδεση. Ο κανονισμός προβλέπει διαδικασίες προκειμένου να συμπεριληφθούν ρήτερη διασφάλιση και μηχανισμοί κατά της στρατη... της τη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και της ΕΚΑΧ και των δύο χωρών. Θα γίνει παρουσίαση πρώτα για τη Μολδαβία και μετά για τη Γεωργία από τους συζητητές μας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Μία παρατήρηση σε ό,τι αφορά την ρήτρα διασφάλισης και το μηχανισμό κατά τη στρατη... καταστρατήγησης που προβλέπει προσωρινή αναστολή δασμολογικών προτιμήσεων. Την περασμένη Δευτέρα συνεδρίασε η Επιτροπή ΑΦΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και συζήτησε εκτενώς την κατάσταση στη Μολδαβία. Παρουσία μάλιστα του Προέδρου του Κοινοβουλίου της Μολδαβίας. Ο Πρόεδρος μας είπε ότι η Μολδαβία θα πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές της ώστε να ξεπεράσει την κρίση που διανύει αυτή τη στιγμή, που έχει κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό χαρακτήρα. Και θα πρέπει να εφαρμόσει τις μεταρρυθμίσεις για να βελτιώσει την οικονομική και κοινωνική κατάσταση της χώρας, κυρίως ε, τις μεταρρυθμίσεις στο δικαστικό σύστημα και την καταπολέμηση της διαφθοράς. Γιατί έχει επιβραδυθεί ο ρυθμός των μεταρρυθμίσεων και της πρόοδου. Μία αναγκαιότητα που επισημάνθηκε και από άλλου συναδέλφου τη ΑΘΕΤ είναι η ανάγκη αύξηση συνεργασία μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων τη Μολδαβία, προκειμένου να υλοποιηθεί αυτός ο στόχος της επιτάχυσης των μεταρρυθμίσεων. Και μάλιστα η εφαρμογή αυτή τη εισβάθος και εκτεταμένη συμφωνία, στα πλαίσια τη συμφωνία σύνδεση θα πρέπει να αποτελέσει τμήμα αυτών των προσπαθειών. Δηλαδή και οι δύο συμβαλόμενε πλευρέ θα πρέπει να εξετάσουν τις συνέπειες ε, αυτών των μεταρρυθμίσεων και πώς θα επηρεάσουν την οικονομία προς όφελος των πολιτών, των νέων κυρίως, ε, τη δημιουργίας θέσεων Απασχόληση και ούτω καθεξής. Και χθε την ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προσέγγιση της Επιτροπής της ε, Πολιτικής Γειτονίας τονίστηκε ότι θα πρέπει και εμείς ε, να βρούμε νέους τρόπους για να βελτιώσουμε την οικονομική και κοινωνική κατάσταση στις γειτονικές χώρες προκειμένου ε. να αυξήσουμε την, προκειμένου να αποτρέψουμε την περαιτέρω αύξηση της έντασης και των πιέσεων και στα κράτη-μέλη. Η συμφωνία σύνδεσης με τη Μολδαβία, όπως οι περισσότερες εμπορικές μας συμφωνίες, περιλαμβάνει και τη ρήτρα διασφάλισης που προβλέπει ότι επιτρέπεται προσωρινή αναστολή των δοσμολογικών προτιμήσεων σε περίπτωση που έχουμε μεγάλη και δικαιολόγητη αύξηση ε, των, εξαγωγών που προκαλεί, μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο στην οικονομία της χώρας εισαγωγής. Οπότε η ρήτρα διασφάλισης αποτελεί τμήμα του γενικότερου πακέτου που σας ανέφερα. Επιπλέον η συμφωνία περιλαμβάνει και το μηχανισμό κατά της στρατε... καταστρατήγησης που προβλέπει δυνατότητα επαναφορά τη ρήτρα του πλέον ευνοωμένου κράτου για την εισαγωγή κάποιων γεωργικών προϊόντων από τη Μολδαβία που ξεπερνούν συγκεκριμένο κατόφλι και μάλιστα χωρί δέους αιτιολόγηση τη προέλευσή του. Με βάση τον κανονισμό του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου, χρειάζεται αντίστοιχη σχετική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να εφαρμοστεί ο σχετικός μηχανισμός κατά της, και της ρήτρας διασφάλισης. Ο προτινόμενος κανονισμός ε, θεσπίζει τις κατάλληλες διατάξεις ε, της Συμφωνίας Σύνδεσης για τις οποίες συμφωνήσαμε ήδη από τον Νοέμβριο του 2014. Η έγκριση του προτινόμενου κανονισμού είναι απαραίτητη για να ε, ενισχυθεί η υποχρέωση της Μολδαβίας που απορρέει από τη συμφωνία και να προστατεύσει τους ε, παραγωγούς όπου χρειάζεται. Η πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπής στηρίζεται κυρίως σε εφαρμογή, συγκρίσιμη εφαρμογή του κανονισμού που ε, έχουν εφαρμοστεί σε συμφωνίες με την Νότια Κορέα, την Κεντρική Αμερική, την Κολομβία και το Περού. Γίνεται μια συγκριτική μελέτης εφαρμογής αυτού του μηχανισμού κατά της καταστρατήγησης και της ρήτρας διασφάλισης και στόχο έχει την εξασφάλιση της οικονομικής ανάπτυξης και εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και ε, στις χώρες της σύνδεσης. Επίσης χαίρομαι για την υποχρέωση υποβολή έκθεσης που έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέναντι στου συναμοθέτης με την δημοσίευση ετήσια έκθεση ε, για την εφαρμογή αυτού του κανονισμού καθώς και του εμπορικού σκέλου της ε, Συμφωνίας Σύνδεσης, γιατί κάτι τέτοιο ενισχύει τη διαφάνεια και την ε, δημοκρατική λογοδοσία σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του κανονισμού. Επίση, εξασφαλίζει το κοινοβουλευτικό έλεγχο τη εμπορική πολιτική τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εξασφαλίζει και πάλι διαφάνεια σε αυτή την εμπορική πολιτική. Και μάλιστα από χθε έχουμε και το σχέδιο πρόταση του Συμβουλίου για το ίδιο θέμα. Οπότε και τα δύο σκέλη τη νομοθετική εξουσία επιταχύνουν τις εργασίες τους. Και δεδομένης και της γνωμοδότησης της Επιτροπής Γεωργίας του Οκτωβρίου, προτείνω στη δική μου έκθεση την έγκριση της πρώτης Ευρωπαϊκής Επιτροπής χωρίς περαιτέρω τροπολογίες. Ελπίζω να συμφωνήσετε με την προσέγγιση μου και περιμένω τις απόψεις για το σχέδιο εξασίσμου, μου, ευχαριστώντας ταυτόχρονα τη Γραμματεία, την Τατιάνα, κυρίως για τη βοήθειά της και τι πληροφορίε που μας έδωσε η Επιτροπή Παρακολούθησης, η Ομάδα Παρακολούθηση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τώρα για τη Γεωργία, ο κύριος Λαντσμπέργκη. Ε, Υπάρχει μια δήλωση του κύριου Βίνκλερ που είναι σκιώδη για τη Μολδαβία. Να σα το διαβάσω τώρα, να σας τη διαβάσω τώρα, χωρί μικρόφωνο. Καλά, τότε καλά. Δεν έχω και πολλά να πω μετά από αυτά που μας είπε ο κύριος Σόλτς δύο θέματα μόνο που ξεχωρίζουν, διαχωρίζουν τη γεωργία από τις υπόλοιπες συνδεδεμένες χώρες που έχουν <clears throat> υπογράψει τις συμφωνίες GFTA. Η Γεωργία είναι η χώρα που έχει κάνει την περισσότερη πρόοδο. Δεύτερον, ο γεωργιανός λαός είναι ο πιο φιλοευρωπαϊκός λαός σε ολόκληρο ε, τον αριθμό των χωρών της ανατολικής γειτονίας και εταιρικής σχέσης. Άρα αυτό είναι πολύ σημαντικό, πρέπει να δώσουμε και εμείς τη σημασία που πρέπει να δείξουμε ότι τους ευχαριστούμε και εκτιμούμε ιδιαίτερα τις προσπάθειές τους και την αφοσίωσή τους. Φυσικά την ρήτρα για την οποία μιλήσαμε κατά της περικύκλωσης νομίζω ότι δεν θα χρειαστεί ε? νομίζω ότι δεν θα χρειαστεί γιατί δεν θα υπάρξει τέτοιος κίνδυνος στο μέλλον και γι' αυτό προτείνω στο σχέδιο ψηφίσματος να μην γίνουν δεκτές σχετικές τροπολογίες Ελπίζω να το δεχτείτε και αναμένω απόψεις. Ευχαριστούμε. Ο Σκιώδης του ΕΛΚ για τη Μολδαβία. Πάλι. Πρόεδρε, συνάδελφοι, ο Σκιώδης δέχομαι την πρόταση της Κομισιόν να εγκριθεί δεσμευτικά η ρήτρα αντικαταστρατήγησης δεν είναι τίποτα καινούριο. Έχει συμπεριληφθεί και στις εμπορικές συμφωνίες της Ένωσης με την Κορέα και την Κολομβία. Όλες οι πτυχές των κανόνων και κανονισμών πρέπει να γίνονται εκτές και από τις δύο πλευρές. Ο σκιώδης του ΕΛΚ θα ήθελα να τονίσω επίσης ότι το Ευρωπαϊκό Κενοβούλιο δέχτηκε την περσινή συμφωνία σύνδεσης με τη Μολδαβία με τεράστια πλειοψηφία. Χαίρομαι γιατί διατηρούμε εδώ την ορμή μας και την ειλικρίνειά μας και αυτό δεν θα έπρεπε να σταματήσει στο επίπεδο της DCFTA. Ελπίζω να συνεχιστούν και οι μεταρρυθμίσεις με το σωστό ρυθμό η Ένωση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ιδιαίτερα θα έπρεπε να υποστηρίξουν όσο περισσότερο μπορούν την προσπάθεια αυτήν. Τώρα, θα ήθελα να εκφράσω την ελπίδα μου να βοηθήσουμε τον εισηγητή με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Uh, Σα ευχαριστώ. Σε ό,τι αφορά τη Μολδαβία θα δώσω το λόγο στον αρχείο των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Σόλτ για τη δουλειά που έκανε και ήδη ε, ο εισηγητή ανέφερε ότι η πρόταση υποστηρίζει διάφορες ε, τοποθετήσει και του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σε ό,τι αφορά τις ε, συμφωνίε που ισχύουν με την Νότια Κορέα, την τα κτλ. Και έτσι λοιπόν έχουν αυξηθεί, έχουν δει πλασιαστεί, μη σας πω και σε κάποια προϊόντα οι εξαγωγές ε, από την ε, Μολδαβία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι εξαγωγές ε, από την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν παραμείνει σταθερές. Το εμπόριο λοιπόν αποτελεί ένα πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο για να υπάρξει και να υποστηριχθεί η μεταρρύθμιση. Το αποτέλεσμα είναι λοιπόν ικανοποιητικό και γι' αυτό λοιπόν είμαι ικανοποιημένο με την απόφαση του εισηγητή για να μην κατατεθούν τροπολογίε στην αρχική πρόταση τη ε, Επιτροπή. Είναι ικανοποιητικό λοιπόν το αποτέλεσμα και αυτό ισχύει και για τα χρονικά όρια. Επίσης, η περίοδος που προβλέπεται για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει τα πράγματα αυτά να κινηθούν γρήγορα, καθώς και η υποχρέωση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δικαιολογεί τα μέτρα τα οποία λαμβάνει. Καλωσορίζουμε λοιπόν την έκθεση του συναδέλφου Σόλτ, καθώ και την υποχρέωση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταθέτει αιτήσια έκθεση προ το Κοινοβούλιο για να υπάρχει δημοκρατικό έλεγχο για την εφαρμογή του κανονισμού αυτού. Θα θέλαμε οι πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις να μην υποσκάψουν τις κοινωνικές και οικονομικές εξέλιξει στη χώρα και νομίζουμε ότι θα πρέπει να υποστηρίξουμε τις προσπάθειες και τις μεταρρυθμίσεις που γίνονται στη χώρα. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον κύριο Σόλτς και ελπίζω να είναι εύκολη η υποστήριξη και η ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο. Να υπάρχει μια ευρεία υποστήριξη. Μάλιστα, λέει ο πρόεδρο, δεν βλέπω από το ECR και από τους πρασίνους να υπάρχει και ότι Δεν ξέρω αν θέλει κάποιο το λόγο να του αντικαταστήσει, να περάσουμε στη Γεωργία. Ο Νίκολα θα μιλήσει για τους σοσιαλιστές και δημοκράτες εξ ονόματος του Σκιωδή. Έχω μια δήλωση από τον συνάδελφο Μόιζε που είναι ο σκιώδης ηγητής για τη Γεωργία και μου ανέθεσε να σας διαβάσω το εξής κείμενο. Είναι υπέρ της πρότασης ε, του κ. Λαντσμπέργκη, δηλαδή να, να γίνει δεκτή χωρί αλλαγέ η πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ό,τι αφορά την εφαρμογή του μηχανισμού κατά της καταστρατήγηση και στη συμφωνία με τη Γεωργία, στη συμφωνία σύνδεση. Και θα πρέπει να εφαρμοστούν οι διατάξεις της ισχύωσης συμφωνίας. Ο κύριος Σόλτ είναι και σκιώδης για τη Γεωργία, οπότε το δίνω το λόγο. Ο Πατρίκ Λιαρίκ, που είναι ο σκιώδη ηγετής για το θέμα αυτό, μου ανέθεσε να σα διαβιβάσω τη γνώμη του. Τονίζει λοιπόν ο κ. Λιαρίκ ότι ανεξάρτητα από την κατάσταση της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Γεωργία, που κατά τη γνώμη του θα μπορούσε να είναι λόγος για να επαναθεωρήσει ή να εξετάσει αναστολή η Ευρωπαϊκή Ένωση του συνόλου της ε, Συμφωνίας Σύνδεσης. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις διατάξεις αυτές και του μηχανισμού είναι σωστή. Η ΓΚΟΕ συμφωνεί με τον εισηγητή ε, να κάνουμε δεκτή την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα πρέπει βέβαια να γίνει μια αξιολόγηση της εφαρμογής του μηχανισμού κατά της καταστρατήγησης, προκειμένου να εφαρμόζεται με καλό επίπεδο αυτοματισμού και να μην επαναληφθεί το φαινόμενο των υπερβολικών ε, εξαγωγών ε, μπανανών από το Περού ή αντίστοιχε περιπτώσει που είχαμε σε συμφωνία με τι Ηνωμένε Πολιτείε. Μια και δεν βλέπω άλλου ομιλητέ, θα δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που είναι ο κ. ο προϊστάμενος της ε, Γενικής Διεύθυνσης για τις έρευνες στην, στο εμπόριο, Φαντάζομαι θα χαίρετε για την ε, θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά το έργο των εισηγητών και των σκιωδών εισηγητών, καθώ και τις γραμματείες τη Επιτροπή σα, και σα ε, ε, επενεί και σας θαυμάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ταχεία διεκπαιρέωση των δύο θεμάτων. Μάλιστα για να γίνει η διεκπαιρέωση στο δυνατόν συντομότερα δεν θα χρειαστούν καν τριμερείς διάλογοι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ολοκληρώσαμε λοιπόν αυτά τα δύο θέματα, την κοινή συζήτηση για τα δύο αυτά θέματα. Να μην ξεχάσουμε την προθεσμία για τις τροπολογίες. 23 Νοεμβρίου, 12 το μεσημέρι, λίγη προθεσμία για τις τροπολογίες. Οπότε κανονικά θα έπρεπε να περάσουμε στο σημείο 7 τώρα, αλλά όπως και εγώ το πρωί έχει κολλήσει στην κυκλοφορία ο Η εισηγήτρια Οπότε περιμένουμε να καταφτάσει μια πολύ σύντομη διακοπή. Okay, colleagues. Thank you. Συνάδελφοι. Έχουμε όλοι προβλήματα κοινωνία, αλλά φροντίστε να έρχεστε εγκαίρως για τα θέματα. Λοιπόν, το επόμενο θέμα είναι το τα. Η σύσταση του 10 για τα κοινωνικά πρότυπα κλπ. Όπως θα θυμάστε το 10 είχαμε εγκρίνει τρεις εκθέσεις ιδίας πρωτοβουλίας από την ίντα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και κοινωνικά και περιβαλλοντολογικά πρότυπα στις εμπορικές συμφωνίες και άλλα. Στο πλαίσιο πάντα των κλιματολογικών αλλαγών και της αντιμετώπισης τους καθώς και για την ανταλλαγή βελτίστων πρακτικών, για τη βελτίωση του γενικότερου πλαισίου όπου μπορεί να γίνει η κοινοβουλευτική επιτήρηση και εποπτεία. Και η συνέχεια που θέλει να δώσει η Κομισιόν πριν κάνει νέες προτάσεις στην έκθεση. Σήμερα έχουμε την πρώτη ανταλλαγή απόψεων λοιπόν για αυτή την καινούργια έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας. Εισηγητής είναι ο κ. Φερέντζη από την ΧΟΕ. Grazie Presidente. eh, anche io voglio iniziare sottolineando... Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ξεκινήσω. όπω είπατε και εσεί ε, τονίζοντα την ε, ανάγκη αυτή. Για πρώτη φορά λοιπόν ε, καλούμαστε να εξετάσουμε πώ τα διάφορα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από το έτος 2010 επηρεάζουν διάφορα θέματα ανθρώπινων δικαιωμάτων και κοινωνική ευθύνη των ε, ε, επιχειρήσεων τη κοινωνική εταιρική ευθύνη. Ξέρουμε τι διάφορε συζητήσει που γίνονται για τη νέα εμπορική στρατηγική τη Ευρωπαϊκή Ένωση, η συζήτηση που διεξάγεται για το TTIP, η μεταρρύθμιση του ΠΟΕ, COP21 στο Παρίσι. Όλα αυτά λοιπόν οδηγούν σε μια νέα μορφή διεθνού εμπορίου ενδεχομένω. και είναι σημαντικό λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να εκφράσει την ε, θέση της. Πιστεύουμε ότι το εμπόριο δεν είναι μόνο η διακίνηση προϊόντων. Επηρεάζει τον 21ο αιώνα και την ζωή των ανθρώπων, την ε, παραγωγικά μοντέλα, γιατί αν προσπαθήσουμε μόνο να πετύχουμε κέρδος, ιδιαίτερα στον χρηματοοικονομικό τομέα, βλέπουμε ότι έχουν σχηματιστεί και έχουν διαμορφωθεί καταστάσει ανταγωνισμού σε ό,τι αφορά τις εργασιακές συνθήκες. Και αυτό ε, πλήττει τα ανθρώπινα δικαιώματα, ε, προκειμένου μόνο και μόνο να υπάρχει κέρδος. Υπάρχουν επίσης ε, περιφέρειες που δεν ασχολούνται ούτε με τα ανθρώπινα δικαιώματα, ιδιαίτερα ούτε με τα περιβαλλοντικά ζητήματα. Γι' αυτό ήθελα λοιπόν να επιβεβαιώσω εδώ κάτι το οποίο αναφέρεται και στην έκθεση ΣΑΕΦΗ. Θα πρέπει να βρεθεί μια ισορροπία μεταξύ των εμπορικών ε, στρατηγικών και των ε, βασικών θεμελιωδών δικαιωμάτων. Το Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να αφήσει τα εργασιακά ζητήματα να ε, έρθουν σε δεύτερη μοίρα μετά τα συμφέροντα των επενδυτών. Ούτε μπορούμε να θεωρήσουμε ότι το ελεύθερο εμπόριο είναι πιο σημαντικό από το περιβάλλον και από τα εργασιακά δικαιώματα. Γι' αυτό λοιπόν προτείνω δύο προτεραιότητες εδώ πέρα. Η μεταρρύθμιση του ΠΟ το 2010 λοιπόν αυτό επιβεβαιώθηκε και το ΠΟ, ο ΠΟ θα πρέπει να μπει στο επίκεντρο των διαφόρων μεταρρυθμίσεων σε ό,τι αφορά και την προβολή των περιβαλλοντικών προτύπων και της ε, ε, των εργασιακών συνθήκων. Και έτσι λοιπόν στο Ναϊρόμπι με τη συμμετοχή του ΠΟΕ και τη ε, Διεθνού Οργάνωση Εργασία θα πρέπει όλα αυτά να προωθηθούν. Τα ανθρώπινα δικαιώματα λοιπόν θα πρέπει να εξεταστούν σε συνάρτηση και με άλλες ε, αρχέ, όπως η αρχή της πλέον ευνοούμενης χώρας. Κάτι άλλο τώρα. Οι διμερείς συμφωνίες είναι σημαντικό να, αξιολογηθούν, ε, να αξιολογηθεί ο αντίκτυπος των ρητρών ανθρωπινών δικαιωμάτων που αποτελούν σημαντικό τμήμα της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά παράλληλα αυτά χρήσουν περαιτέρω βελτίωση. Θα πρέπει λοιπόν από εκείνου να αναλογιστούμε το πώς μπορούν να διαμορφωθούν με πιο αποτελεσματικό τρόπο σε ό,τι αφορά τη διαδικασία προσφυγών, για παράδειγμα δυνατότητα προσφυγής ε, που θα πρέπει να αφορά και να δίδεται ως δικαίωμα και σε ενώσεις τοπικές, όχι μόνο σε ΜΚΟ. Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να εκτελεστούν στο έπακρο. Τα ανθρώπινα δικαιώματα λοιπόν και η άσκηση τους, η εφαρμογή τους είναι αξιόπιστη μόνο όταν υπάρχει ανεξαρτησία και θα πρέπει επίσης να υπάρχουν και σχετικοί δείκτες. Θα πρέπει επίσης να διευρυνθούν αυτοί οι δείκτες, να υπάρχουν και άλλα κριτήρια, όπως για παράδειγμα η ηλικία, το φύλλο και όλα αυτά είναι σημαντικά. Αυτό το έργο θα το συνεχίσουμε και σε συνάρτηση με την ομάδα Gender Mainstreaming για την ε, ενσωμάτωση της διάστασης των φύλων σε όλα τα ζητήματα αυτά και ευχαριστώ όλους με τους οποίους συνεργάστηκα. Είναι πάρα πολύ σημαντική η συζήτηση και επίσης υπήρξε και μια σχετική μελέτη η οποία εξέτασε την εμπορική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με την άρτηση του φύλου Επίση, σε ό,τι αφορά του επενδυτές, προτείνεται το θέματα να το εξετάσουμε και σε συνάρτηση και με τα θέματα ανεργία. Ο ειδικό εισηγητή από πλευρά του Κοινοβουλίου τόνισε ότι τα κοινωνικά δικαιώματα θα πρέπει να έχουν προτεραιότητα όταν υπάρχει θέμα σύγκρουση με του επένδυτες. Επίσης ε, και στις ε, συμφωνίε θα πρέπει να υπάρχουν διάφορα κοινωνικά κριτήρια, όπω η πρόσφαση των γυναικών, των παιδιών και άλλα τέτοια ζητήματα, τα οποία συχνά παραμελούνται και τα αναπαραγωγικά δικαιώματα είναι σημαντικά. Οι αλλαγέ ε, του κλίματο και όλοι αυτοί οι παράγοντε φυσικά είναι όλο και πιο σημαντικοί. Θα πρέπει λοιπόν να εξασφαλίσουμε ότι τα... οι προσυπογράφοντες στη συνθήκη των ΗΠΑ θα εφαρμόζουν τα πρότυπα αυτά το ζήτημα του περιορισμού της αύξησης της θερμοκρασίας σε 2 βαθμούς Κελσίου. Θα πρέπει να αναλογιστούμε εκ νέου το ρόλο τον οποίο μπορούν να δραματίσουν οι διεθνείς συμβάσεις, γιατί θα πρέπει να εξετάσουμε τις σχετικές ρήτρες για το περιβάλλον ε, στον δρόμο προς το COP21 και στα προβλήματα τα οποία ενδεχομένω θα προκύψουν θα πρέπει να είμαστε ενωτόμη σε ό,τι αφορά τις εμπορικές συμφωνίες και τον αντίκτυπο των οποίων ενδεχομένω έχουν σε θέματα εκπομπών. Και αυτό ασφαλώς θα είναι ουσιώδους σημασία τα επόμενα χρόνια, αν θέλουμε να υπάρχει και αντίκτυπο των συμφωνιών της COP21. Ένα άλλο ζήτημα είναι η εταιρική ευθύνη η κοινωνική εταιρική ευθύνη. Είναι κάτι το οποίο εξετάζουμε από το 2012 ως ένα σύμφωνο μεταξύ των πολιτών και των εταιριών. Είναι ένα μεγάλο βήμα προς τα εμπρός, αλλά θα πρέπει να δούμε ότι και οι επενδύσεις θα πρέπει πάντα να λαμβάνουν υπόψη και τις ε, κοινωνικές συνέπειες. Επίσης, να λαμβάνουν υπόψη και τα θεμελιώδη δικαιώματα των ατόμων και των ε, τα ζητήματα αυτά όμως της κοινωνικής ευθύνης δεν ξέρω κατά πόσο ε, λαμβάνουμε επαρκή προσοχή σε ό,τι αφορά και την ε, ε, διεθνοποίηση των εταιριών. και την παγκοσμιοποίηση των εταιριών. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να είναι πολύ πιο δεσμευτικός ο σεβασμός των κοινωνικών αυτών δικαιωμάτων. Και το τονίζω ότι οι κοινωνικές ρήτρες ε, στις, εταιρικές, ε, στις εμπορικές συμφωνίες συχνά δεν ε, τυχάνουν του απαραίτητου σεβασμού και χρειαζόμαστε τις απαραίτητες εγγύησεις για να είναι πραγματικά δεσμευτικές οι ρήτρε κοινωνικής ευθύνη των εταιριών. Κοιτώντα και τις ιδέες του Εκβαδόρ, της Νοτιού Αφρική για τα θέματα αυτά, θα πρέπει να τους δώσουμε τον απαραίτητο σεβασμό και να διασφαλίσουμε ότι γίνονται πάντα εξάντε αναλύσεις ε, και μελέτες τύπου πρωτού υπογραφούν οι εμπορικές συμφωνίες. Γι' αυτό λοιπόν ζητούμε και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προωθήσουν ε, τις πρωτοβουλίες σε ό,τι αφορά την κοινωνική ευθύνη, σε ό,τι αφορά την εξαγωγή και την όρεξη ε, μεταλλαγμάτων. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να κοιτάξουμε και θέματα ορεικτού πλούτου. Υπάρχει το θέμα των στρατιωτών, των παιδιών στρατιωτών, των ε, ματωμένων διαμαντιών και το καθεξής. Θα πρέπει επίσης, ε, Πρόεδρε, να αναφέρουμε δύο βασικές προκλήσεις. Καταρχάς το εύρος όλων των ζητημάτων τα οποία προσπάθησα να καλύψω και αυτό το διευκρινίζω και στην εισαγωγή μου. Και κατά δεύτερον, είναι η πρώτη φορά που η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου έχει καθήκον να εξετάσει και τις εκθέσεις που στο παρελθόν έχει εγκρίνει η το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να προσπαθήσει να βρει κατευθυντήρε γραμμέ. Θα πρέπει να βρούμε μια μεθοδολογία σε ό,τι αφορά και τι μελέτε τύπου Και ελπίζω αυτό να καταστεί κάτι το μόνιμο σε ό,τι αφορά την ΙΝΤΑ, την Επιτροπή τη Εμπορίου και θεωρούμε ότι μπορούμε να συμβάλλουμε και να δώσουμε σημαντικές συστάσεις και για το Κοινοβούλιο και για την Επιτροπή και για τις ε, διαπραγματεύσει για τις εμπορικές συμφωνίες. Θα ήθελα να υπάρξει μια έκθεση βάση πραγματικών αποτεκτικών στοιχείων. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω του συναδέλφου και τους κοιόδης εισηγητέ που έχουν συνεργαστεί μαζί μου έω τώρα, καθώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που μα βοηθάει και συνεργάζονται ιδιαίτερα επικοδομητικά μαζί μα. Ελπίζουμε να μπορέσουμε να Έχουμε τη τελική ανάλυση ένα κείμενο πολύ χρήσιμο για το μέλλον του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Εκτενή παρουσίαση. Όταν όμω διαβάζετε ε, κείμενο γραπτό, προσπαθήστε να το διαβάζετε με κάπως αργό ρυθμό για να σας προλαβαίνουν και οι διερμηνεί. Θα ακούσουμε τώρα τα σχόλια των σχεδόν εισηγητών. Πρώτα, η σχεδόν εισηγήτρια του ΕΛΚ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, η έκθεση αυτή θα μα επιτρέψει να κάνουμε έναν απολογισμό των συστάσεών μα του 2010 και μάλιστα ήμουν εισηγήτρια για τα ανθρώπινα δικαιώματα και του κοινωνικού και περιβαλλοντικού κανόνε των διεθνών εμπορικών συμφωνιών, όπω είπε και η εισηγήτριά μα η κυρία Φορέντσα. Πιστεύω ακραδαντά ότι οι κοινωνικοί και οι περιβαλλοντικοί κανόνες και τα εμπορικά συμφέροντα μπορούν να ενισχυθούν παράλληλα εφόσον ε, όλες οι χώρες και όλοι οι συντελεστές εφαρμόζουν τους ίδιους κανόνες. Έχουμε πολυμερείς διαλόγους και εμπορικές διαπραγματεύσεις ε, με κεφάλαιο αηφόρο ανάπτυξη ε, στι διμερεί μα σχέσει. Γι' αυτό θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στην ουσιαστική εφαρμογή των εμπορικών συμφωνιών. Φαίνεται ότι το παρόν πλαίσιο είναι ε, βέλτιστο για την έκθεση αυτή. Βέβαια, στα πλαίσια της μεταρρύθμισης του SPZ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ε, υποβάλει έκθεση για την εφαρμογή του ενισχυμένου συστήματος δασμολογικών προτιμήσεων. Σε ό,τι αφορά το ΕΡΕΣ, ε, πριν από δύο χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε το Παγκόσμιο Σύμφωνο για την Αηφορία. Μετά την τραγωδία του εργοστασίου Ραναπλάτσα στο Μπαγκλαντές. Οπότε είναι ενδιαφέρον να εγκύψουμε και στο σημείο αυτό. Σε ό,τι αφορά τους περιβαλλοντικούς κανόνες, και εδώ είχαμε εξελίξεις μετά το 2010 με την έναρξη των εμπορικών διαπραγματεύσεων σε ό,τι αφορά τα φιλοπεριβαλλοντικά αγαθά και τις τεχνολογίες και περιμένουμε ανυπομονησία και τις εργασίες της COP21 για να δούμε ε, αν ε, θα επιτευχθεί η συμφωνία για το κλίμα και πώς θα εμπεριλάβει τις εμπορικές πτυχές. Όπως και η κυρία Φλωρέντσα, ελπίζουμε να γίνει μια σωστή και φιλόδοξη ερμηνεία και εξελόγηση της εφαρμογής των συστάσεων το 2010. Κέρκεντελ, σκιώδη συγγήτρια των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών κολλείεται δυστυχώς. Μου ζήτησε όμως ε, να παρουσιάσω εγώ τις απόψεις της ε, θα ακολουθήσω τη συμβουλή που έδωσα πριν και θα προσπαθήσω να διαβάσω αργά τις σημειώσεις. Ε, είναι ευκαιρία με, την έκθεση αυτή να κάνω μια αξιολόγηση του προγράμματος που τέθηκε πριν από 10 χρόνια. Ε, ζητήσαμε για παράδειγμα συνδυασμό των περιβαλλοντικών κοινωνικών προδιαγραφών και των προδιαγραφών για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε όλες τις ε, εμπορικές, ε, διμερείς εμπορικές συμφωνίες και τις διεθνείς συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην παρακολούθηση της εφαρμογής αυτών των δικαιωμάτων και προδιαγραφών με τακτική ενημέρωση και υποβολή εξέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των συμβαλωμένων χωρών προς την κοινωνία των πολιτών και ζητεί ανοιχτή διαδικασία με συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων και επανεξέταση της συμφωνίας για την επίλυση των διαφορών. Επίσης, ε, σε ό,τι αφορά το σύστημα ε, γενικευμένων προτιμήσεων, ζητούμε αναστολή το, του, του καθεστώτος αυτού σε περίπτωση που εντοπίζεται παραβίαση. Επίση, το θέμα τη κοινωνική εταιρική ευθύνη ε, χρήζει διευκρίνηση ε, και αποκατάσταση απο, αποτελεσματικότητα και συμπερίληψη σε όλε τι εμπορικέ συμφωνίε, ε, ακόμη και σε αυτέ για, το, για τι δεσμολογικέ προτιμήσει. Επίση, ζητούμε από τι επιχειρήσει υποχρεωτικά να υποβάλουν τον απολογισμό του RCU. Σε σχέση με τις, ε, με τις θέσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής χαιρόμαστε που έλαβε υπόψη τις συστάσεις μας, παρόλο που δυστυχώς ε, η πραγματικότητα δεν ανταποκρίνεται στις συστάσεις. Για παράδειγμα, ε, στη, στην συμφωνία με την Κορέα είχαμε υποβάθμιση των προδιαγραφών μας. Σε ό,τι αφορά τη συμφωνία του ελπίζουμε να υπάρχει φιλόδοξο περιβαλλοντικό κεφάλαιο, αν και φαίνεται ότι θα είναι από τα λιγότερα φιλόδοξα τελικά που έχει διαπραγματευτεί ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν εξασφαλίζεται ούτε σωστή παρακολούθηση, ούτε σωστή εφαρμογή των ούτως ή άλλως ε, άτολμων ε, δεσμεύσεων. Σε ό,τι αφορά τις συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης με τη Δυτική Αφρική, οι προδιαγραφές είναι ακόμη χαμηλότερες. Σε ό,τι αφορά το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων, θα πρέπει να δούμε τις σχέσεις μας με τη Γουατεμάλα και τη Σοζιλάνδη. Εκεί γίνεται κατάφορη και συστηματική παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Απόδειξη ότι το σύστημά μας δεν λειτουργεί. Ό,τι αφορά την ευθύνη για την αλυσίδα ανεφοδιασμού, το πρόβλημα το εντοπίσαμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν από μία πενταετία. Και πολλοί μη κρατικοί παράγοντες ε, δεν χρησιμοποιούν ε, το CSR με αποτέλεσμα να έχουμε σοβαρέ παραβιάσεις. Ελπίζω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αγγίψει τα θέματα αυτά και να προτείνει λύσει. Θα πρέπει να εμπνευστούμε από προηγούμενε επιτυχεί ε, εμπειρίες, όπω ε, την βελτίωση τη πυρασφάλεια των Μπαγκλαντέ μετά το ατύχημα στο εργοστάσιο Ράνα Πλάσα. Ε, θα πρέπει να γίνει μια ενημέρωση και επικαιροποίηση των συστάσεων του 2010. Βέβαια, είναι γνωστή η απροθυμία του Συμβουλίου να αναλάβει δράσει για παραβιάσει. Σε ό,τι αφορά τη συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους και εκπροσώπους κοινωνίας των πολιτών. Θα μπορούσαμε να προσκαλούμε εκπροσώπους ε, ε, των ομάδων αυτών στις ε, ομάδες παρακολούθησης Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θέλουμε να συμβάλλουμε με επικοδομητικό τρόπο στην έκθεση αυτή και να συνεργαστούμε με τις πολιτικές ομάδες για τη διεκπαιρέωση αυτού του σημαντικού έργου. Αυτά από το σκία της ηγετρία των σοσιαλιστών. Και τώρα θα δώσω το λόγο στη Μαρία Ντεσσαρνές που είναι η σκιώδη συγγήτρια των φιλελευθέρων. Oh, sure. Ah, sorry. Okay. Α, ah, λάθος, λάθος. Ευχαριστώ. Μπερδεύτηκα προς το για λίγο. Δεν άκουσα την ε, πρώτη εισήγηση, αλλά η ομάδα μου και εγώ προσωπικά με χαρά δεχόμαστε το ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παραμένει στην πρωτοβουλία των εκκλήσεων για μια πιο αποτελεσματική σύνδεση μεταξύ εμπορίου και αξιών που πρέπει να ενισχυθούν όπως το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, βιώσιμη ανάπτυξη, σεβασμό του περιβάλλοντος και προστασία αυτού καθώς και την κοινωνική προστασία. Είναι καλό ότι αυτά, αυτές οι αξίες ε, τονίζονται περισσότερο στις διμερείς συμφωνίες μέσα στο γενικότερο σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων πρέπει να παίζουμε όντως ηγετικό ρόλο γιατί έτσι μπορούμε να έχουμε αποτελέσματα με τις εταίρες μας και το ίδιο να κάνουμε και με τις Ηνωμένες Πολιτείες και με τις Αφρικανικές χώρες και άλλες. Υπάρχουν και άλλα θεματι... άλλες θεματικές ή οριζόντιες εκθέσεις όπως τα ορυκτά από χώρες σειράξεων κλπ. Όπως σας είπα η ομάδα μου είναι δεσμευμένη στην ενδυνάμωση των αξιών αυτών και μέσω του εμπορίου. Αλλά αυτά βέβαια δεν μπορούν να μετρηθούν και να αποτιμηθούν παρά μακροπρόθεσμα. Παρ' όλα αυτά πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ό,τι εργαλεία διαθέτουμε για την ενδυνάμωση αυτών των καθολικών αξιών στις οποίες πιστεύουμε, αλλά ταυτόχρονα είμαστε ρεαλιστές, διότι δεν μπορεί μόνο το εμπόριο να καταλήξει στην εφαρμογή και χρήση αυτών των αξιών, αλλά χρειάζεται μια ευρύτερη ε, εξωτερική πολιτική της Ένωσης με περισσότερες διπλωματικές προσπάθειες κλπ. Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε αλλά να μην έχουμε και την αυταπάτη ότι μόνο η εμπορική πολιτική μόνη τη θα λύσει τα προβλήματα που έχουμε στον σύγχρονο κόσμο. Ευχαριστούμε, συγγνώμη που σας μπέρτεψα. Η πράσινη τώρα, η Σκά Κέλλερ. Ευχαριστώ πολύ. Πράγματι το εμπόριο δεν είναι το μόνο εργαλείο, αλλά είναι ένα από τα εργαλεία, νομίζω συμφωνούμε όλοι. Και αυτό πρέπει να το λέμε πάντοτε και στις εκθέσεις μας για να παρατηρούμε και πώς το εφαρμόζουν οι υπόλοιποι. Ακόμα χρειάζονται πολλά βέβαια για τη σύνδεση ανθρωπίνων δικαιωμάτων με εμπόριο ας πούμε πρέπει να γίνουν ακόμη πολλά. Επίσης οι όροι που θέτουμε τι εμπορικέ συμφωνίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα θα μπορούσαν να ενισχυθούν αλλά και να καταδικάζουμε όσους δεν τους εφαρμόζουν με βάση τις αρχές της συνέπειας της πολιτικής μας, της νεκτικότητας. Όσο για τα θέματα εμπορίου και βιώσιμης ανάπτυξης, η έκθεση συνιστά τη συμπερίληψη μιας δεσμευτικής ρήτρας αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα εφαρμόζεται κιόλα. Αυτό πρέπει ακόμη να το επεξεργαστούμε. Πρέπει οι όροι που θέτουμε να είναι και εφαρμόσιμοι και να ενδυναμώσουμε τον εποπτικό μηχανισμό ο οποίος είναι μέχρι τώρα αναποτελεσματικός και να καλέσουμε την Κομισιόν να εφαρμόσει και περισσότερες κυρώσεις. Επίσης πάλι για τα ανθρώπινα δικαιώματα ανέφεραν ήδη οι συνάδελφοι το θέμα της αξιολόγησης για βιώσιμη ανάπτυξη πριν από τις ε, διαπραγματεύσεις αλλά και μετά είναι σημαντικό και πρέπει στις εκθέσεις μας να συμπεριλαμβάνουμε και αξιολογήσεις για το σεβασμό των ανθρωπινών δικαιωμάτων όπως έχει, έχουν πει και άλλοι να γίνεται αποτίμηση της αξιολόγησης και ως προς τις συμφωνίες για τα τρόφιμα Είχε πει το Κοινοβούλιο ότι θέλει από τη στρατηγική του 10 ήδη να συμπεριληφθούν τέτοιες αρχές. Δεν έγινε τίποτα τέτοιο, αλλά ούτε και στη νέα στρατηγική. Αυτό πρέπει να το τονίσουμε. Έχουμε δει και μερικές καταστροφές ως προς τις συνθήκες εργασίας, ιδιαίτερα στην υφαντουργία. Πρέπει να το παρακολουθήσουμε και αυτό, όλα πρέπει να τα παρακολουθήσουμε. Και να έχουμε τις κατευθυντήριες γραμμές για τα επιχειρήσεις ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα υποχρεωτικές και δεσμευτικές. Και για την εφαντουργία και για άλλους τομείς. Υπάρχει σαφής ανάγκη να νομοθετήσει η Ένωση για αυτό το θέμα. Αυτό πιστεύουμε εμείς. Τώρα εμπόριο και κλίμα. Εδώ έγιναν μερικές σημαντικές συστάσεις που εμείς οι πράσινοι συνυπογράφουμε και τώρα. Μεταρρύθμιση του ΠΟΕ για να γίνεται διαχωρισμός των προϊόντων και ως προς την μεταποιητική μέθοδο και την προέλευση και τονίζουμε ότι οι υποχρεώσεις και οι στόχοι που προβλέπονται από ισχύουσες συνθήκες και με τον ΟΗΕ πρέπει να έχουν προτεραιότητα έναντι οποιασδήποτε στενότερης ερμηνείας και να δημιουργηθεί μια παγκόσμια οργάνωση περιβάλλοντος. Ο αθέμητος ανταγωνισμός, δηλαδή το dumping, είναι επίσης ένα άλλο πρόβλημα και για τη μεταρρύθμιση της ETS. Τελευταία ζητήσαμε καλύτερη προσαρμογή και για τις εκπομπές διοξιδίου. Και τέλος, το 10 ήδη μιλούσαμε για το κόστος που, έχει επί του περιβάλλοντος, που έχουν επί του περιβάλλοντος οι μεταφορές των προϊόντων. Και, αυτό, και σε αυτό δίνουμε ιδιαίτερη σημασία. Νομίζουμε ότι δεν πρέπει να επεκταθεί η σημασία αυτών των μεταφορών διότι παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο, έχουν μεγάλο μερίδιο στις κλιματολογικές αλλαγές. Επιλεκτικά σας τα είπα και συνοπτικά, αλλά αυτά θέλουμε να τονίσουμε εμείς ως ομάδα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ και τώρα θα ήθελα να ακούσουμε την εκπρόσωπο του EFTD. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Φορέντσα για την εξαιρετική δουλειά που έκανε το θέμα των περιβαλλοντικών προτύπων, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τη εταιρική κοινωνική ευθύνη και τη ε, εμπορική πολιτική και η αλληλοσύνδεση όλων αυτών είναι κάτι που μα απασχολεί ιδιαίτερα. Και θα ήθελα και εγώ να σα αναφέρω ότι σε θέματα ε, επιχειρήσεων είμαι πολύ υπέρ τη εταιρική κοινωνική ευθύνη. Είμαστε πραγματικά ε, υποστηρίζουμε την έννοια αυτά και η εργασία της Επιτροπής Επασχόλησης ήταν πάρα πολύ καλή και ελπίζουμε ότι η συγγετρία θα λάβει υπόψη την γνωμοδότηση της Επιτροπής αυτής και πρέπει να σας πω ότι η συγγετρία της γνωμοδότησης σε ό,τι αφορά τη σημασία της Συμφωνίας ILO και των Διεθνών Συμβάσεων θα πρέπει αυτά να αποτελούν κίνητρο για την ένταξη στην συνθήκη της, του ILO. Και νομίζω ότι αυτό είναι λοιπόν σημαντικό για μια εμπορική πολιτική που θα τηρεί και θα προωθεί τις βασικές αξίες. Το ελεύθερο εμπόριο και οι σχετικές συμφωνίες θα πρέπει να υποστηρίζουν την ανάπτυξη περιβαλλοντικών προτύπων και θα πρέπει να υπάρχουν κυρώσεις για όσους δεν σέφονται τους ε, σχετικούς κανόνες. Και επίσης καλό θα ήταν να υπάρχουν, ε, δεν είναι νόημα έχει να υπάρχουν ad hoc δικαστήρια, αλλά να μην υπάρχουν κυρώσεις για όσους παραβιάσουν τις διτάξεις Κατανοώ επίση το ρόλο των ε, μελετών ε, περιβαλλοντικού αντικτύπου. Θεωρώ ότι θα πρέπει να γίνονται και πριν και μετά τις διαπραγματεύσεις τέτοιες εκθέσεις, αλλά προφανώς η πιο σημαντική φάση είναι πριν την επικύρωση. Και συμφωνώ με την ε, έκκληση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναπτύξει νέα στρατηγική για την εταιρική κοινωνική ευθύνη. Και διαρκώς επαναλαμβάνουμε ότι προτού αλλάξει η νομοθεσία πρέπει πρώτα να αλλάξει η κουλτούρα που επικρατεί. Ελπίζω λοιπόν να λάβετε υπόψη την γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και ελπίζω να συνεργαστούμε ενεργά. Ευχαριστώ, ο Πρόεδρος. Έχουμε λίγο χρονική πίεση και θα πρέπει να πάμε λίγο πιο γρήγορα. Έχουμε τρεις ομιλητές. Σας παρακαλώ να, είμαστε, να είστε σύντομοι η κυρία Ρένα, η ε, Κομισιόν και μετά η Θήτρια. Ευχαριστώ, Ντέιβιτ. Πολύ γρήγορα. Συμφωνώ με τα περισσότερα σχόλια που ακούσαμε και ευχαριστώ την κυρία Φορέντσα για το έργο της και την παρουσίαση που μας έκανε γιατί στάθηκε στις ε, βασικότερες αρχές ό,τι αφορά το σεβασμό των ανθρωπίνων, ε, κοινωνικών και περιβαλλοντικών δικαιωμάτων. Για τους σοσιαλιστές τρεις είναι οι βασικές προτεραιότητες που θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο έγγραφο και οι περισσότερες έχουν ήδη συμπεριληφθεί. Πρώτον, δεσμευτική ε, διάταξη, γιατί το να επαφιόμαστε στην καλή προαίρεση δεν αρκεί θα πρέπει να έχουμε δεσμευτική εφαρμογή των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και ανθρώπινων δικαιωμάτων. Επίση, η διαδικασίε παρακολούθηση με ταυτόχρονο μηχανισμό επιβολή κυρώσεων. Και επίση, άσχετα με τα οικονομικά συμφέροντα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κοινωνικά, περιβαλλοντικά και ανθρώπινα δικαιώματα θα πρέπει να υπερισχύουν, να αποτελούν προτεραιότητα και να μην ισχύουν διπλά μέτρα και σταθμά ανάλογα με το ποιο είναι ο συνομιλητή μα. Ευχαριστώ ευχαριστώ και τώρα ο κύριο Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είμαι συντονιστή και εκπροσωπώ την ομάδα τη Ευρώπη των Εθνών και των Ελευθεριών. Αυτό που μπορούμε να πούμε για την έκθεση είναι ότι ναι, μεν, η υπερθέρμανση του πλανήτη θα πρέπει να καταπολεμηθεί, αλλά έχει κόστο ε, αυτή η καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών και το να ζητήσουμε από τα κράτη-μέλη επενδύσεις ε, για την ενεργειακή μετάβαση πρέπει να έχουμε υπόψη ότι θα κοστίσει 7 δισεκατομμύρια ευρώ. Και αυτό για το εμπορικό ισοζύγιο των κρατών μελών ε, θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα. Δεν μπορούμε να του τα επιβάλλουμε λοιπόν υποχρεωτικά. Και σίγουρα η λογική των οικονομικών και των εμπορικών συμφωνιών δεν θα πρέπει να συνδέεται με τα ανθρώπινα δικαιώματα, γιατί θα πρέπει επιθετικά να εξαγάγουμε τις αξίες μας σε άλλα ως λαούς που ίσως ε, αισθανθούν ε, ότι τους υπαγορεύουμε πράγματα επιθετικά. Θα πρέπει να σεβόμαστε την εθνική κυριαρχία. Επίσης, η δική μας αντίληψη για τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν μπορεί να επιβάλλεται στο όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Θα πρέπει ε, ε, να έχουμε μια σχέση μεταξύ περιβαλλοντικών και εμπορικών συμφωνιών. Αλλά το ότι ε, θέλουμε οπωσδήποτε να βρούμε τέτοιου δεσμούς δεν θα πρέπει να μας οδηγήσει σε υπερβολική γραφειοκρατία. Η δημιουργία ενός παγκόσμιου οργανισμού περιβάλλοντος έχει κάποιο νόημα, αλλά δεν θα πρέπει να γίνει υπερεθνικός αυτός ο οργανισμός και να μην ε, υπερέχει έναντι των εθνικών κρατών, για να μην ε, υποβαθμίσει την αρχή της εθνικής κυριαρχίας. Ευχαριστώ. Η κυρία Σίλβια Φερμεντίνη είναι η συντονίστρια πολιτικών στην Γενική Διεύθυνση Εμπορίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα είμαι λακωνική μια και μας πιέζει ο χρόνος κύριε Πρόεδρε και όπως ακούσαμε η συζήτηση είναι πραγματικά ευρύτατη και απαιτείται πολλής χρόνος για να επισέλθουμε σε όλες τις πτυχές. Πάντως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά το ζωηρό ενδιαφέρον της Επιτροπής σας ε, για μια αηφόρο πολιτική εμπορική που θα λαμβάνει υπόψη και την ανάπτυξη και θα υφετήσουμε και στο μέλλον αυτή την προσέγγιση. Είχαμε πολλές διεθνείς εξέλιξεις από το 2010, γι' αυτό και είναι πολύ επίκαιρη η στιγμή αυτή του υπολογισμού, του απολογισμού συγγνώμη, προκειμένου να χαράξουμε και τη μελλοντική μας στρατηγική. Ε, και στι αρχέ του έτου μάλιστα έχουν εγκριθεί και νέοι αναπτυξιακοί στόχοι. Είχαμε εξελίξει ε, και στι δράσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αναφέρθηκαν ε, σε αυτό οι προλαλήσαντε. Ε, όλο και περισσότερο χρησιμοποιούμε ε, στι διμερεί εμπορικέ συμφωνίε και ρήτρε βιώσιμη ανάπτυξη. Επίση, έχουμε τη μεταρρυθμίση του συστήματο γενικευμένων προτιμήσεων ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά του δικαιούχου του νέου συστήματο, του ενισχυμένου για τι γενικευμένε εκτιμήσεις. Αναφέρθηκε το θέμα των συμφωνιών με το Μπαγκλαντές, με την ε, Μιανμάρ. Συμμετέχουμε σχετική πρωτοβουλία για τα εργασιακά δικαιώματα στο Μιανμάρ. Και έχουμε ξεκινήσει να προωθούμε δυναμικά σε όλα τα διεθνή φόρα το θέμα της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης. Τέλος, να αναφερθούμε στις βασικές εξελίξεις της αξιολογής που κάνουμε. Πολύ σημαντικό αυτό. Θα πρέπει να είμαστε συνεκτικοί και να έχουμε μελέτη επιπτώσεων κάθε φορά που προτείνουμε την έναρξη νέων διαπραγματεύσεων και θα πρέπει να μην ξεχνούμε τη διάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πρόσφατα είχαμε και καταθυντήριες γραμμές ε, για τη λήψη υπόψη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη μελέτη επιπτώσεων των εμπορικών μας πολιτικών. Αυτό το έργο είναι δυναμικό εξελικτικό και ήδη έχουμε σημαντική πρόοδο. Τέλος, ήθελα να πω ότι η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί το επίκεντρο και της εμπορικής μας πολιτικής ε, και τώρα και για το μέλλον και είναι σαφής η ε, δέσμευσή μας υπέρ μιας διαφανούς και βιώσιμης ε, εμπορικής πολιτικής. Είναι σημαντική η συνοχή και η συνέπεια η εφαρμογή των μηχανισμών που έχουμε είναι απαραίτητη και η εφαρμογή των κεφαλαίων ανάπτυξη, ε, βιώσιμης ανάπτυξης στις εμπορικές μας συμφωνίες είναι πολύ σημαντικό, αλλά κάτι τέτοιο προποθέτει τη συνοχή των διαφόρων πολιτικών, την ευθυγράμμιση των εμπορικών πολιτικών με τις αναπτυξιακές πολιτικές. Έτσι θα μπορέσουμε να εφαρμόσουμε και εμπράκτος μεταρρυθμίσεις στις συμβαλόμενες μας χώρες και στις χώρες εταίρου. Επαναλαμβάνω, χαίρομαι για το ενδιαφέρον σας για το θέμα αυτό και θα συνεχίσουμε τις συνομιλίες με την Επιτροπή σας και μέσω των συναντήσεων που θα έχουμε με την εισηγήτρια και τους σκιώδεις εισηγητές. Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ για τη λακωνικότητά σας. Όπως είπατε θα επανέλθουμε στο θέμα αυτό και άλλη στιγμή. Και τώρα, εν συντομία, το λόγο στην εισηγήτρια για να ολοκληρώσουμε το θέμα αυτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομη. Θα ήθελα απλώς να πω ότι από την πρώτη αυτή ανταλλαγή απόψεων διαπιστώνω μια μεγάλη σύγκληση και συνένεση mm. ως προς τις προτεραιότητες και τους μηχανισμούς στους οποίους θα έπρεπε να επικεντρωθεί η έκθεση. Διαπιστώσαμε την αδυναμία των κοινωνικών ρητρών και την ανάγκη μεγαλύτερης παρακολούθησης των πιο δεσμευτικών ρητρών, καθώς και την ανάγκη πρόβλεψη ενός μηχανισμού επιβολή κυρώσεων. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλου τους, και και τους συναδέλφους που έλαβαν το λόγο και θεωρώ ότι με συνεργασία θα καταλήξουμε σε μια καλή έκθεση. Θα συνεννοηθώ με τους σκιώδεις ηγητές για την επόμενη μας συνάντηση ήταν πραγματικά πολύ σημαντική συμβολή των συναδέλφων και θα λάβω υπόψη τα σχόλιά του στην περαιτέρω διαμόρφωση της έκθεσής μου. Σας ευχαριστώ. Σίγουρα θα συνεδριάσουν οι σκιώδεις με την εισηγήτρια. Εμείς στις 25 Ιανουαρίου θα εξετάσουμε την ε, έκθεση αυτή και στις 8 Φεβρουαρίου 12 το μεσημέρι θα λήξει η προθεσμία ε, για την υποβολή τροπολογιών. 13 και 14 Μαρτίου κατά πάσα πιθανότητα θα ψηφίσουμε και κατόπιν θα περάσει την Ολομέλεια. Περνάμε τώρα στις ψηφοφορίες. Ελπίζω να έχετε φέρει και τις ε, ηλεκτρονικές κάρτες ψηφοφορίας. Θα ψηφίσουμε καταρχήν την ετήσια έκθεση για την ΕΤΕ για το 2014. Ο Γιάννη Ζαντό είναι ο εισηγητής μας. Οι τροπολογίες 1 και 9 έχουν αποσυρθεί. Ψηφίζουμε τροπολογία 2. Ποιο είναι υπέρ. Α, συγγνώμη, έχουμε συμβαστική τροπολογία 1. Mm. Αυτή καλύπτει τι τροπολογίε 1 και 9. Ποιο είναι υπέρ τη συμβαστική τροπολογία 1. Κατά. Εγκρίνεται. Και περνάμε στην τροπολογία 2 που είναι συμβατή με τη συμβαστική. Ποιο είναι υπέρ, κατά, Αποχέ. εγκρίνεται. Τροπολογία 3 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 2. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 8 καταπίπτει. Τροπολογία 7 το ίδιο. Και πάμε στη συμβαστική 3. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Μάλλον απορρίπτεται, αλλά στο ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Συμβαστική τροπολογία 3 παρακαλώ. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Αν ψηφίσετε όλοι, λίγη η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Δεκατέσσερις ψήφοι υπέρ, 20 κατά. Μία αποχή. Απορρίπτεται με σαφή διαφορά. Περνάμε τώρα στη βαστική 4. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 23 αποσύρεται. 13 και 14 καταπίπτουν. Τροπολογία 16 απαρά, μη παραδεκτή. Η 18 καταπίπτει. Οπότε πάμε στη συμβαστική 5. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 20. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 21 υπέρ. Α, θέλετε ηλεκτρονικό έλεγχο. Για την τροπολογία 20 λοιπόν ηλεκτρονικός έλεγχος άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος, εγκρίνεται με 22 ψήφους υπέρ και 13 κατά. Τροπολογία 21, ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται με την ίδια διαφορά. 22 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 24 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 26 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται 27 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 28 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 30 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 31 υπέρ Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 31. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. 18 υπέρ, 17 κατά. Εγκρίνεται. 32 υπέρ. Κάτα. Νομίζω ότι η ίδια είναι η πλειοψηφία, αλλά θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ και το 32 έναρξη. Για την 32. Πέρας. 18 υπέρ, 17 κατά, εγκρίνεται. 33 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 37 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 38 υπέρ. Κατά. Αποχές έγκρινεται. 39 υπέρ. Κατά. Αποχές έγκρινεται. 40 υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά ας το ελέγξουμε. 40, 40. Η 40. 6 υπέρ, 12 κατά, 17 απόχες, απορρίπτεται. 41 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 42 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 43 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 44 υπέρ. Σε τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά.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 32 υπέρ. Κανείς κατά. Δύο αποχές. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στον Γιάννεκ. Ωραία. Ετήσια έκθεση για την πολιτική στρατηγική ανταγωνιστικότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 5. Υπέρ. Κατά. απόχέ, απορρίπτεται. Η 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές Ας ελέγξουμε παρακαλώ την 7. Ηλεκτρονικά. Πέρα. 17 υπέρ, 18 κατά. Αυτή απορρέπεται λοιπόν με μια ψήφο διαφορά. Συμβασική 2 υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται. Τροπολογία 10 υπέρ. Κατά. Ας αλλάξουμε παρακαλώ και την 10. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρας. 16 υπέρ, 19 κατά, απορρίπτεται. Η 11 υπέρ. Κατά. Αποχές, απορρίπτεται. Η 12 υπέρ. Κατά. Αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 14 υπέρ. Κατά. Ας ελέγξουμε παρακαλώ το 14. Νομίζω ότι έχει απορριφθεί, αλλά για να είμαστε σίγουροι ας ψηφίσουμε ηλεκτρονικά το 14. Πέρας της ψηφορίας. Με σαφή διάφορα. 11 υπέρ, 22 κατά, απορρίπτεται. Τροπολογία 15 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές έγκρινεται. Τροπολογία 18 υπέρ κατά αποχές έγκρινεται. Η 19 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές έγκρινεται. Η 22 υπέρ κατά αποχές Νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά θα ελέγξουμε την 22 παρακαλώ. Πέρας. 20 υπέρ, 13 κατά, εγκρίνεται 23 υπέρ. Κατά. Νομίζω ότι και αυτή θα πρέπει να την ελέγξουμε. Για την 23 παρακαλώ ψηφίζουμε. Πέρας. 15 υπέρ, 19 κατά μία αποχή, απορρίπτεται. 24 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 6 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 27 υπέρ. Α, συγγνώμη, καταπίπτει. Συμβαστική 7 υπέρ. 28, λέει ο πρόεδρο. Ναι, συγγνώμη, συγγνώμη. 28 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβαστική 7 υπέρ. Κατά. Αποχές έγκρινεται. Και η τροπολογία 32 τώρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές έγκρινεται. Τελική ψηφοφορία. Έναρξη ηλεκτρονικής ψηφοφορία, παρακαλώ. Πέρασε. 30 υπέρ, 3 κατά, 2 αποχές εγκρίνεται και συγχαρητήρια στον εισηγητή. Και έχουμε και άλλη μία. Άλλη δύο. Επόμενη ψηφοφορία για έναρξη διαπραγματεύσεων με Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία προφορική ερώτηση. Ποιο είναι υπέρ τη προφορική ερώτηση. Έχουμε και μια τροπολογία του κ. Κάσπαρη για την παράγραφο 7. Ποιο είναι υπέρ της προσθήκη Κατά αποχές εγκρίνεται. Και για το σύνολο της προφορικής ερώτησης. Ποιος είναι υπέρ. Ηλεκτρονικά θα ψηφίσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας εγκρίνεται με 30 ψήφους υπέρ και 4 κατά. Εγκρίνεται λοιπόν. Και ψηφίζουμε για την έναρξη των διαπραγματεύσεων ε, του τριμερούς διαλόγου έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων και τα εμπόρια ορισμένων αντικειμένων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν χρειάζονται τουλάχιστον 21 ε, ψήφοι για να εγκρίνουμε την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων. Προκειμένου να καταλήξουμε σε συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση. Οι τροπολογίες έκθεση ε, υιοθετήθηκαν στις 27 Οκτωβρίου στην Ολομέλεια και έγινε αναπομπή στην ε, Επιτροπή. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία, άρχιτη ψηφοφορία. Πρέπει να το διαβάσω για τα πρακτικά. Η προτινόμενη απόφαση προβλέπει την έναρξη επίσημων διοργανικών διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο και την Επιτροπή προκειμένου να, φτάσουμε, να καταλήξουμε συμφωνία με πρώτη ανάγνωση. Οι τροπολογίε που εγκρίθηκαν στι 27 Οκτωβρίου θα αποτελέσουν τη βάση τη διαπραγματευτική εντολή που απαρτίζεται ε, και τη διαπραγματευτική ομάδα που απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον εισηγητή και του και εισηγητέ. Άρχεται ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Και αν ψήφισατε όλοι λίγοι η ψηφοφορία, 34 ψήφοι υπέρ, χωρί καμία αρνητική ψήφο και μία αποχή. Εγκρίνεται λοιπόν η έναρξη των διοργανικών διαπραγματεύσεων και ολοκληρώσαμε και τι ηλεκτρονικέ μα ψηφοφορίε. Θα περάσουμε τώρα στο σημείο 12, την εφαρμογή και επανεξέταση της Στρατηγικής Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Κεντρική Ασία. Έκθεση πρωτοβουλίας. Έγινε ήδη η πρώτη ανταλλαγή απόψεων στις 26 Οκτωβρίου. Σήμερα θα συζητήσουμε το θέμα της στρατηγικής με εκπροσώπους των χωρών και επιχειρηματιών. Ο εισηγητής ο κ. Μπορέλη δυστυχώς απουσιάζει, αλλά τον αντικαθιστά ο Ντάριο Ταμπουράνο. Κύριε Ταμπουράνο, αναπληρώνω τον κύριο Μπορέλη, οπότε έχετε και το λόγο. Al collega Borrelli a leggere il suo δεν είναι παρόν ο εισηγητής γιατί έχει αρνηλημένες υποχρεώσεις στο εξωτερικό. Η πρόταση γνωμοδότηση για την θεώρηση στρατηγική για τις χώρες της Κεντρικής Ασία θα ήθελε λέει να επαναλάβει ορισμένες από τις έννοιες που πρότεινε ο εισηγητής. Η Κεντρική Ασία είναι μια στρατηγική πρόκληση που ξεπερνάει κατά πολύ το μόνο Αφγανιστάν και που δικαίως ή αδίκως ε, μα επέσυρε την προσοχή μας. Η Ευρώπη που καθορίστηκε από το 2008 χρήζει τροποποίηση η Ευρωπαϊκή Στρατηγική. Το πρότυπο περιφερειακής ανάπτυξης ε, Ευρώπης, Ασίας και τα λοιπά και η διαδικασία της Σαγκάης. Και επίσης άλλαξαν οι ενεργειακές επενδύσεις των Ηνωμένων Πολιτειών εκεί. Αυτό είναι το γενικότερο πλαίσιο τη γνωμοδότηση και περνάω κατευθείαν στο πρώτο σημείο. Η γνωμοδότηση βασίζεται σε τρεις άξονες. Ο πρώτο είναι η ενδυνάμωση των εμπορικών σχέσεων και συναλλαγών, ημερών συναλλαγών με τη χρήση των υπαρχουσών συνθήκων με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ώστε να υπάρξει ενισχυμένη συνεργασία και τερκή σχέση όπως έγινε και με το Καζαχιστάν. Δεύτερος άξον εσωτερικές δομικές μεταρρυθμίσεις για να δημιουργηθεί θετικό εμπορικό κλίμα για τις ε, ξένες επενδύσεις. Τρίτος άξον πολιτική στήριξη στις δραστηριότητες confidence building μεταξύ των χωρών της ε, περιοχής. Είναι ουσιώδες να ενισχυθεί η θέση της Ένωσης στην Ασία για να αναπτυχθούν οι διμερείς εμπορικές σχέσεις και συναλλαγές. Όσο για τις τελευταίες αυτές με την Ευρώπη, προς στιγμή βασίζονται κυρίως στο Καζαχστάν που είναι στατικός εταίρος της Ένωσης. Πρέπει όμως να διευρυνθούν οι δραστηριότητες αυτές και, και προς άλλες χώρες για να παρασπιστούμε καλύτερα τα εμπορικά μας συμφέροντα διεθνώς. Η αποτελμάτωση με το Τουρκμενιστάν είναι χαρακτηριστική. Το είδαμε την τελευταία ε, ομάδα που συνεδρίασε για την πρόοδο των σχέσεων αυτών. Το Τουρκμενιστάν πρέπει να θεωρηθεί και αυτό ο στρατηγικός εταίρο για τη σταθεροποίηση της περιοχής γενικότερα. Και αυτά τα λέει στο σημείο 2. Στο σημείο, στα σημεία 3 και 4 γίνονται πιο συγκεκριμένε προτάσει για τι εμπορικέ σχέσει. Η Κεντρική Ασία είναι μια ζώνη στρατηγικά σημαντική και ω προ την ενέργεια και ω προ τη διαφοροποίηση των ενεργειακών μα πηγών. Και πολλέ ευρωπαϊκέ επιχειρήσει είναι ήδη δραστηριε εκεί και επομένω η Ένωση πρέπει να ενισχύσει τη διαφοροποίηση των οικονομιών τη κεντρική Ασία που χρειάζεται επενδύσει σε νέε τεχνολογίε, βιώσιμη ανάπτυξη κλπ. και τηλεπικοινωνίε και επικοινωνίε στο σημείο 5 γίνεται λόγος για την εσωτερική διαρθρωτική μεταρρύθμιση, για μεγαλύτερη εσωτερική ανάπτυξη ξένες επενδύσεις και αυτό σημαίνει ενίσχυση του κράτους δικαίου, μείωση των διοικητικού άχθους, καταπολέμηση της διαφθοράς, αναμεταρρύθμιση της δικαιοσύνη και δημιουργία θετικού περιβάλλοντος για τις επενδύσεις. Τέλος, το σημείο 6 είναι πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό αυτό το σημείο 6. Η Ευρώπη πρέπει να βοηθήσει την περιοχή αυτή στον εκδημοκρατισμό της και τον εξυγχρονισμό της, αλλά πολλά θα εξαρτηθούν από το κατά πόσο θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε κλίμα εμπιστοσύνη μεταξύ των χωρών της περιοχής. Εδώ υπάρχουν πολλοί φραγμοί για τη δημιουργία ενός τέτοιου κλίματος εμπιστοσύνης. Υπάρχουν ακόμη εθνοτικές διαφορές και διαμάχες και σειράξεις και ο ρόλος της παιδείας εδώ μπορεί να είναι πολύ σημαντικός. Είμαστε πεπισμένοι ότι οι χώρες αυτές πρέπει να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Erasmus Συν. Είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει μια προσπάθεια συνεργασίας και συνέργειας να δημιουργήσει μια νέα δηματική για την ε, συνεργασία μεταξύ των χωρών αυτών διαμεθοριακή συνεργασία που λέμε στην ΑΦΕΤ ή στην ΕΠΕΞ φάνηκε ότι πρέπει η Ένωση να παίξει σημαντικότερο ρόλο εκεί και το ζητούν εξάλλου αυτό και οι χώρες της περιοχής. Τα φορά τεχνογνωσίας και εμπορικής ανάπτυξη περιφερειακή. Πρέπει βέβαια να υπάρχουν όπως είπα και πριν ε, σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ ημών και εκείνων οι χώρες της Κεντρικής Ασίας θέλουν να ενδυναμώσουν το διάλογο και τις ανταλλαγές και συναλλαγές τους με την Ένωση παρά την ύπαρξη ορισμένων δυσκολιών και διαφωνιών. Πρέπει λοιπόν να έχουμε μια διαφοροποιημένη προσέγγιση αναχώρα. Πρέπει να στείλουμε ένα σαφές μήνυμα προς τους στρατηγικούς αυτούς μας εταίρους και αυτό πόσο μάλλον τώρα που υπάρχει αποσταθεροποίηση σε χώρες που είναι κοντά στην περιοχή αυτή. Ευχαριστώ πολύ και αναμένω με αδειμονία τις ε, συμβολές σας. Εκτός μικροφώνου, Πρόεδρος. Όπισε for e Να ακούσουμε από το ΕΛΚΑ. Ευχαριστώ και ευχαριστώ και τον εισηγητή για την έκθεσή του. Έχω μερικά σχόλια. Πιστεύω ότι δεν αρκεί να λέμε ότι η Κεντρική Ασία είναι περιοχή γεωστρατηγικής σημασίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί αυτή την ορολογία τη χρησιμοποιούμε στη σχέση μας με την ευρύτερη περιοχή. Και η προηγούμενη στρατηγική, παρόλο που είχε αυτή την ορολογία, δεν ήταν και πολύ επιτυχημένη και αποτελεσματική. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επένδυε σε προγράμματα υποδομής ε, στην ενέργεια και προσπαθούσε να ασκήσει πίεση στις κυβερνήσεις για να σεβαστούν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αλλά η πίεση δεν απέδωσε, γιατί δεν είχαμε φαίνεται αρκετά μέσα και χρησιμοποίησαν οι κυβερνήσει αυτέ τα κοινωτικά κονδύλια για να χρηματοδοτήσουν τι υποδομέ του και τα δικά του τα εθνικά κονδύλια τα χρησιμοποιούσαν για την αύξηση τη ασφάλεια και την ενίσχυση των ε, στρατιωτικών του ικανοτήτων. Οπότε χρησιμοποίησαν τα δικά μας κονδύλια ε, για να κάνουν δική τους δουλειά, κάτι που θα έπρεπε να την είχαν αναλάβει οι ίδιοι. Τώρα προσπαθούμε με μια νέα στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αλλάξουμε κάπως την προσέγγιση μας στο θέμα αυτό. Δύο είναι οι βασικοί στόχοι. Το πρώτο στόχος είναι να επαιδείουμε στο ανθρώπινο δυναμικό, στον κόσμο. Και αυτό δεν το αναλύουμε αρκετά. Δεν μιλούμε επαρκώς για την ε, ενίσχυση αυτού του πυλώνα. Και επίσης ε, ε, χρηματοδότηση προγραμμάτων για την ανάπτυξη των ανθρώπων, των κατοίκων της περιοχής αυτής. Επίσης θα πρέπει να επαναφέρουμε αυτές τις χώρες της Κεντρικής Ασίας στο διεθνές σύστημα ελεύθερων συναλλαγών. Γιατί οι μεγάλες χώρες γύρω από την Κεντρική Ασία, η Ρωσία δηλαδή και η Κίνα, έχουν σημαντική παρουσία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μόνο τρίτη ή τέταρτη σε σημασία παράγων περίπτωση τέταρτο σημασία παράγων. Οπότε θα πρέπει να επαναφέρουμε τι χώρε αυτέ στο διεθνέ σύστημα ε, ελεύθερων συναλλαγών και να τι προσελκύσουμε σε αυτέ τι παγκόσμιε σχέσει. Θα πρέπει να συνδυάσουμε λοιπόν τι επενδύσει στο ανθρώπινο δυναμικό με τι υπόλοιπε επενδύσει, τροποποιώντα κάπω τη στρατηγική μα. Επαναλαμβάνω, η προηγούμενη μα στρατηγική στην Κεντρική Ασία δεν απέδωσε ιδιαίτερου καρπου. Η Μαρία Ρένα είναι η, συγητρία, η σκιώδη συγγήτρια για τους σοσιαλιστές και δημοκράτες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Νταβίτ, ευχαριστώ Νταβίτ Μπορέλη για όλη αυτή τη δουλειά. Δεν συμμερίζομαι απόλυτα την άποψη του συναδέλφου από το ΕΛΚ που λέει ότι υπήρξε πλήρης αποτυχία της στρατηγικής. Πρέπει να προσέξουμε ορισμένα σημεία της που διαφέρουν από χώρα σε χώρα της Κεντρικής Ασίας. Αν συγκρίνουμε ας πούμε το Τουρκμενιστάν με το Ουσμπεκιστάν βλέπουμε ότι οι καταστάσεις είναι τελείως διαφορετικές. Συμφωνώ ότι πρέπει να υπάρξει διαφοροποιημένη προσέγγιση αναχώρα. Πολύ σημαντικά σημεία εξάλλου ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα μας φαίνονται πολύ σημαντικό να τα θίξουμε και αυτά. Έγινε λόγος για την ενεργειακή σημασία της περιοχής αυτής. Σε περιβαλλοντικό επίπεδο βλέπουμε ότι η εκμετάλλευση των ενεργειακών και ορυκτών πόρων δημιουργεί, γίνεται με τρόπο που καταστρέφει πολλές φορές το περιβάλλον και άρα πρέπει εδώ να ενδιαφερθούμε ιδιαίτερα για αυτό το θέμα της περιβαλλοντολογικής ανάπτυξης της περιοχής που θα στηρίξει εξάλλου και τον πληθυσμό. Χρειάζεται εδώ μια ιδιαίτερη προσπάθεια γιατί οι πληθυσμοί αυτοί, οι λαοί αυτοί δεν έχουν δικαιώματα, δεν έχουν πρόσβαση και αυτά όλα τα θίγει η έκθεση του κύριου Βορέλη, καθώς και η καταπολέμηση της διαφθοράς. Μια έκθεση της Κομισιόν δείχνει ότι είναι από τις πρώτες χώρες στη διαφθορά οι χώρες αυτές. Άρα χρειάζεται μια προσπάθεια κατά της διαφθοράς αλλά και υπέρ της ευθύνη των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται εκεί. Πρέπει να ξέρουμε ποιοι είναι ακριβώς οι μηχανισμοί που εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις για να καταπολεμήσουν τη διαφθορά εκεί. Τίθεται και ένα ερώτημα ως προς τη διεύρυνση προς άλλες χώρες. Πρέπει και αυτό να το συζητήσουμε. Χρειάζεται με τη σημερινή κατάσταση της ε, Κεντρικής Ασίας να διευρύνουμε την εταιρική σχέση και σε άλλες χώρες όπως την Μογγολία. Πρέπει να τεθεί μεταξύ των εισηγητών. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα να περάσουμε στην Άλτε. Ο κύριος Στακουλά. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εμείς θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον εισηγητή, ο οποίος ε, έκανε πολύ καλή εκκίνηση στο θέμα αυτό και νομίζω ότι πολλά σωστά σημεία ε, ανέφεραν και οι υπόλοιποι ομιλητές. με πολλά εξ των οποίων πρέπει να πω ότι σύμφωνα. Από πλευρά τη Άλτε θα ήθελα να πω ότι θα πρέπει ε, ασφαλώς και να υποστηρίξουμε και να εμβαθύνουμε τις σχέσεις και ε, τη συνεργασία με τις χώρες αυτές. Και νομίζω ότι πολλούς ε, στόχους έχουμε εκείνους και αυτό ασφαλώς μπορεί να αποτελέσει μια καλή βάση συνεργασία. Αν ε, φυσικά πληρούνται ορισμένοι όροι γιατί στην περίπτωση αυτή θεωρώ ότι μπορούμε να υποστηρίξουμε και την ανάπτυξη της χώρας αυτές και νομίζω ότι πολλά θα μπορούσε να συνεισφέρει ε, βοηθήσει, σε πολλά σημεία θα μπορούσε να βοηθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στι χώρε αυτέ, σε ό,τι αφορά τι υποδομέ, σε ό,τι αφορά την σταθερότητα στι χώρε αυτέ. Σε κάποιε από τι χώρε αυτέ, ωστόσο, πολλά θα πρέπει να γίνουν, πολλοί όροι θα πρέπει να πληρούνται αν θέλουμε να πετύχουμε ένα καθεστώ ελεύθερη αγορά, Οικονομία τη αγορά. Και εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν θα πρέπει να συμβάλλει αυτά που τις αναλογούν. Αυτό που είναι ανησυχητικό είναι η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις χώρες αυτές. Προφανώς η Ευρωπαϊκή Ένωση και εμείς ως ε, βουλευτές της, ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, θεωρούμε ότι ακρογωνία ολίθο το σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πρόκειται για κάτι το οποίο είναι αδιαπραγμάτευτο, αναπαρατρίωτο. Θα πρέπει να αποτελούν αυτά τμήμα των ε, σχέσεων συνεργασία με τι χώρε αυτέ και θα πρέπει να είμαστε ειλικρινεί. Έχουμε προβλήματα σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προφανώ θα πρέπει να κανονίσουμε πρώτα τα του οίκου μα, αν θέλουμε να έχουμε αξιοπιστία ε, ενώπιον των χωρών αυτών. Και αυτό είναι κάτι το οποίο καθημερινά πρέπει να παρακολουθούμε στο ιστορικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορούμε να μιλάμε μόνο στους άλλους για ανθρώπινα δικαιώματα και να μην φροντίσουμε τα εσωτερικά μας. Παρά το γεγονός αυτό, η, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι ένα θέμα το οποίο έχει την αντίστοιχη προσοχή το 2011, επικυρώθηκε και η συμφωνία με το Ουσμπεκιστάν παρά την ανησυχητική κατάσταση που επικρατεί στο Ουσμπεκιστάν σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ένα άλλο σημαντικό σημείο το οποίο θα πρέπει να καταπολεμήσουμε είναι η διαφθορά. Το ανέφεραν άλλωστε και οι συνάδελφοι. Και μπορούμε να υποβοηθήσουμε τις χώρες αυτές στην καταπολέμηση της διαφθοράς. Ας συνεχίσουμε λοιπόν την ενεργή συνεργασία με τις χώρες της Κεντρικής Ασίας και μέσω της συνεργασίας αυτής μπορούμε να βοηθήσουμε λοιπόν τις χώρες να πετύχουν ε, κράτη πιο σταθερά και να ενταχθούν στην ε, παγκόσμια αγορά. Εν συντομία λοιπόν κύριε Πρόεδρε, αυτά είναι, αυτές είναι οι τοποθετήσεις της Άλντε. Σας ευχαριστώ. Εκ μέρους της ΓΚΟΕ, ο κύριος Σόλτς. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Θα συμφωνήσω και εγώ με την κριτική που άσκησε ο προηγούμενος ομιλητής. Αναρωτιόμαστε όμως, υπάρχει πραγματικά κάποια στρατηγική ή μήπω πρόκειται για μια, ένα συνονθήλευμα διαφορετικών μέτρων, διαφορετικών μέσων που σε κάποιε περιπτώσει εφαρμόζονται, σε κάποιε άλλε δεν εφαρμόζονται σε ό,τι αφορά τι χώρε τη Κεντρική Ευρώπη, τη Κεντρική Ασία. Τα παρατήματα από μόνο και ο αριθμό των παρατημάτων μα καταδεικνύουν ότι δεν έχουν ουσιαστικά συμβεί ουσιαστικά πράγματα τα τελευταία χρόνια και πώ θα μπορούσε να διαμορφωθεί μια διαφορετική στρατηγική για να υπάρχει βιώσιμη ανάπτυξη και οικονομία προς όφελος των πολιτών των χωρών αυτών. Όταν βλέπουμε την ε, ανεργία των νέων να φτάνει 80-90% σε κάποιες περιφερειές, αυτό νομίζω ότι καταδεικνύει με σαφήνεια τι είδους προοπτικές μπορεί να έχουν οι νέοι στις χώρες αυτές. Και βλέπουμε λοιπόν ότι είναι παρόμοια η κατάσταση με την κατάσταση που επικρατεί στη Μέση Ανατολή, με όλες τις κοινωνικο-οικονομικές συνέπειες και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι πραγματικά λοιπόν είναι επιτακτική ανάγκη να σκεφτούμε ποια οικονομικά μέσα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την ε, εμπορική πολιτική προκειμένου και να καλυφθεί το χαμένο έδαφος. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να πω ότι ευχαριστώ τον ε, συνάδελφο και τον εισηγητή Μπορέλη για τα σημεία που μας παρουσίασε αλλά καλό θα ήταν να τονιστούν κάποια σημεία παραπάνω για να είναι σαφή η στοχοθέτηση όταν λέμε ότι θέλουμε η Κεντρική Ασία να αποτελεί στρατηγικό εταίρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει παράλληλα να διαπιστώσουμε ότι όπως αναφέρεται στο σημείο 3 πρόκειται για μια τεράστια φιλοδοξία και εδώ θα πρέπει να τονίσουμε ότι δεν πρόκειται μόνο για θέμα διαφοροποίησης των πηγών ενέργειας το οποίο οικονομικά και πολιτικά είναι μεγάλο συμφέρον και μεγάλη ανησυχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά αν θέλουμε όντως να είναι στρατηγικός εταίρος θα πρέπει να κοιτάξουμε πολλά, πολλές άλλες επιτυχίες ε. και αυτό που το Συμβούλιο κατέθεσε ως πόρισμα και ως συμπεράσματα για τη νέα στρατηγική για την Κεντρική Ασία θεωρώ ότι περιλαμβάνει πολλά καλά σημεία, καλή τα κράτη-μέλη να καταβάλουν μεγαλύτερες προσπάθειες για την ε, ενεργειακή συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κεντρικής Ασίας προκειμένου με τον τρόπο αυτό να συμβάλλουν στην σταθερότητα και την ασφάλεια στην ε, περιοχή και αυτό θα πρέπει να ειδωθεί σε συνάρτηση με όσα συζητάμε σήμερα και δεδομένων των όσων συνέβησαν στον ε, Παρίσι. Όσο τραγικά και αν ήταν αυτά τα περιστατικά θα πρέπει να έχουμε την ειλικρίνεια να διαπιστώσουμε και να δούμε ποια ε, εμπορικά εργαλεία πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και προσβλέπω στη συνεργασία με τον ε, εισηγητή προκειμένου να περάσει η γνωμοδότηση. Ευχαριστώ. Εκ μέρους ε, των Πρασίνων τώρα, ο κύριος Βουίκνερ. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο και εγώ ευχαριστώ τον κύριο Μπορέλη για την καλή αυτή έκθεση, η οποία ασφαλώς ε, αποτελεί ένα πάρα πολύ καλό σημείο αφετηρίας για τις εργασίες μας. Με ικανοποιεί η βασική στάση για μια ενισχυμένη εμπορική συνεργασία, αλλά σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα θα ήθελα να πάμε και να δούμε παραπάνω από ότι υπονόησε ο προηγούμενος ομιλητής, ε, γιατί βλέπετε τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν ε, είναι ότι παραβιάζονται τα κράτη αυτά μόνο, αλλά στο Αζερμπαϊτζάν οι εξαγωγές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση προϋποθέτει την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα πρέπει να αλλάξουν οι όροι. Θα πρέπει να επιβληθεί η βάση για μας. Θα θέλουμε να συνάψουμε τις συμφωνίες αυτές, αλλά βάσει κοινών αξιών. Επαναλαμβάνω, η κεντρική αφρικανική περιοχή είναι ύψης της σημασίας για μας προφανώς, αλλά δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα αυτά εις βάρος ε, ατόμων που διώκονται. Ο άνθρωπος είναι πάνω απ' όλα. Ας δούμε το Καζακστάν. Έχουμε ενισχύσει την ε, εμπορική συνεργασία, ωστόσο η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχει επιδεινωθεί. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να ενταχθούν και μηχανισμοί εποπτείας στις ε, συμφωνίες αυτές. Το Ουσπικιστάν, από ό,τι φαίνεται, η συνεργασία με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας και με την ε, κυβέρνηση του Ουσμπεκιστάν έχει βελτιωθεί. Και φαίνεται εξωτερικά λες και έχει καταργηθεί η παιδική εργασία, αλλά ε, στην ουσία δεν έχει καταργηθεί. Άρα θα πρέπει να προσέξουμε τι γίνεται και με τις επίσημες εκθέσεις και η καταναγκαστική εργασία σε κάποιο βαθμό έχει καταργηθεί, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχει καταργηθεί πλήρως. Άρα θα πρέπει να κοιτάξουμε και να ερευνούμε όλες αυτές τις καταστάσεις με μεγαλύτερη προσοχή και στο Τουρκμενιστάν. Τα προβλήματα στην κλωστή φαντουργία εξακολουθούν να είναι πάρα πολύ σημαντικά. Προσβλέπω λοιπόν στην συνεργασία και ελπίζω να μπορέσουμε να πετύχουμε κάτι όχι μόνο για τη δική μας οικονομία στην Ευρώπη αλλά και για τα ανθρώπινα δικαιώματα και για το περιβάλλον στις χώρες αυτές. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν η FTT έχει εκπρόσωπο. Ο κύριος Φερά, ο συντονιστής ε, της ομάδας CNF. Ευχαριστώ. Για τις διεθνείς προκλήσεις και 25 χρόνια μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, ε, ποια είναι η παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κεντρική Ασία. Σίγουρα προσπαθούμε να επέβουμε σε αυτή την σφαίρα επιρροής, παρόλο που είναι έθραυστα τα κράτη. Έχουμε τρεις διαφορετικές ζώνες επιρροής, της Κίνας, της Ρωσίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τα μοντέλα επιρροής ε, της Κίνας και της Ρωσίας είναι ακόμη παρόντα στην Κεντρική Ασία. Γι' αυτό και δυσκολεύεται η Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβάλλει το δικό της μοντέλο, το οικονομικό και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, προκειμένου να τις προσελκύσει σε πιο δημοκρατικά καθεστώτα. Προσοχή όμως ε, για το πώς διαπραγματευόμαστε. Ε, θέλουμε να ενταχθούν το Ουσπεκιστάν και το Τουρκμενιστάν στο Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Πρόκειται όμως για ασταθείς ε, χώρες και ζώνες. Θα πρέπει να είμαστε λοιπόν συνετοί και προσεκτικοί και κυρίως να σεβαστούμε τις άλλες χώρες που έχουν επιρροή στην περιοχή αυτή. Και δεν θα πρέπει της, ε, την ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Αφρικής να τη μετατρέψουμε σε ζώνη αντιπαράθεσης με τη Ρωσία. Ευχαριστώ. Έχουμε τώρα τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Λουκ που είναι προϊστάμενος ε, της αρμόδιας ε, υπηρεσίας Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη σχέση με την Κεντρική Ασία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να σχολιάσω εντάχει τις παρατηρήσεις των Ευρωβουλευτών που αποδεικνύουν ότι η Κεντρική Ασία είναι περιοχή με ιδιαίτερο στρατηγικό ενδιαφέρον για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταρχήν να διευκρινίσουμε το εμπόριο της επενδύσεις και το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κεντρική Ασία. Αυτή τη στιγμή διαδραματίζουμε πολύ σημαντικό ρόλο στις εμπορικές επενδύσεις σε όλες τις χώρες της Κεντρικής Ασίας. Είμαστε από τις πέντε σημαντικότερους εμπορικούς τους εταίρους. Και με τη μεγαλύτερη οικονομία, το Καζακστάν, είμαστε υπαριθμόν ένα εμπορικό εταίρο σε ό,τι αφορά ε, και το εξωτερικό εμπόριο και τις αλλοδαπές επενδύσεις. Και το μισό περισσότερο FDI του Καζακστάν προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις έχουν σημαντική παρουσία εκεί. Βέβαια, η κατάσταση επιδέχεται βελτιώσεις, γι' αυτό είναι σημαντικό να έχουμε περισσότερη συνεργασία με τις χώρες αυτές, όχι μόνο με το Καζακστάν και τις υπόλοιπες χώρες της Κεντρικής αξίας. Και η σημαντική προϋπόθεση γι' αυτό είναι και οι χώρες αυτές να ενταχθούν στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου και να αισθενιστούν τους παγκόσμιου κανόνε του εμπορίου. Είχαμε επιτυχείς εμπειρίες για την τεχνογνωσία που δώσαμε στο Καζακστάν και στο Τατζικιστάν. Το Καζακστάν θα προσχωρήσει ως ο νούπος των ΠΟΕ και, το... και προσπαθήσαμε ε, να παρατηρήσουμε και το Τουρκμενιστάν και το Ουσμπεκιστάν να εισέλθουν. Αν και είναι πιο απρόθυμες αυτές οι χώρες να ενταχθούν στον ΠΟΕ. Σε ό,τι αφορά την ε, διευρυμένη εμπορική σχέση με το Καζακστάν προωθείται και διαρευνούμε και άλλους τρόπους ενισχυμένη συνεργασία με τις υπόλοιπες χώρες της Κεντρικής Ασίας. Γι' αυτό και είναι σημαντική η σχετική συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις προσπάθειές μας να αναβαθμιστούν, σε ό,τι αφορά τα εμπορικά θέματα, χρήσιμο ήταν που ακούσατε προηγουμένως την κυρία Φορμεντίνη που ανακεφαλαίωσε τις προσπάθειες Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για το εμπόριο και την βιώσιμη ανάπτυξη. Στο καθεστώς, ε, το ενισχυμένο καθεστώς ε, γενικευμένων προτιμήσεων έχουμε έτοιμη την πρόταση που θα υποβάλουμε στο εγγύς μέλλον στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με σκοπό να παρακολουθούμε εκ του συνήκη στην εφαρμογή των εργασιακών και των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Και το θέμα του Ουσπικιστάν για την κλωστή φαντουργία είναι πολύ σημαντικό. Συζητήθηκε τον προηγούμενο, την προηγούμενη άνοιξη και θα συνεχιστούν οι συζητήσεις. Επαναλαμβάνω, υπάρχει χώρος για βελτιώσεις, παρόλο που έγινε σημαντική πρόοδος, αν συγκρίνουμε την κατάσταση με το παρελθόν. Είχαμε εντυπωσιακές εξελίξεις, παρόλο που αναμένονται ακόμη περισσότερες και η ΔΟΕ επιβεβαίωσε την πρόοδο των χωρών αυτών. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε ε, τις συνεργασίες των ουσμπικικών αρχών με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας για την μεγαλύτερη εδραίωση των εργασιακών δικαιωμάτων. Σε ό,τι φορά το περιβάλλον, άλλες χώρες έχουν ζωηρότερο ενδιαφέρον και άλλες όχι. Το Καζακστάν, για παράδειγμα, ενεργοποιήθηκε σε περιβαλλοντικά θέματα και η διεθνή έκθεση που θα γίνει στο Καζακστάν του χρόνου θα επικεντρωθεί σε θέματα ενέργεια και αναζήτηση ε, καινοτόμων λύσεων. Έχουμε μάλιστα και κεφάλαιο για τι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια στην ενισχυμένη οικονομική σχέση με το Καζακστάν. Δεν ξέρω αν οι συνάδελφοι από την υπηρεσία εξωτερικών σχέσεων θα ήθελα να πει κάτι για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η κυρία Περκούσιαν θέλει να σχολιάσει κάτι για το ρόλο της ΕΕΤ στις χώρες αυτές. Ναι, θα προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομη. Ένα σημαντικό στοιχείο είναι η εισαγωγή της αρχής της διαφοροποίησης, δηλαδή στοχεύουμε να αντικατοπτρίζουμε την προθυμία των εταίρων μας στην Κεντρική Ασία να διαφοροποιηθούν από τους γείτονές τους. Έχουν διαφορετικές, διαφορετικούς στόχους και θέλουν με διαφορετικό τρόπο να προχωρήσουν τις διμερείς μας σχέσεις. Πρέπει και αυτό να το λάβουμε υπόψη μας. Επίσης θα ήθελα να σημειώσω δύο πρόσφατες εξελίξεις σημαντικές όπως τον ορισμό ενός νέου εκπροσώπου της Ένωσης για την Κεντρική Ασία, τον Πέτρο Μπούριαν, που είναι πολύ ενεργός στην πρόθεση της συνεργασίας και στην ε, δημιουργία στενότερων σχέσεων. Και έπειτα το νέο πολιετές ενδεικτικό πρόγραμμα μέχρι το 2015 15 με 20 που είναι σημαντικό για την ενίσχυση της συνεργασίας μας. Επίσης πρέπει να σημειώσω ότι το κράτος δικαίου, η παιδεία κλπ. έχουν το, τύχει ιδιαίτερη προσοχή στην ενδυνάμωση των σχέσεών μας στους τομείς αυτούς με τις χώρες της Κεντρικής Ασίας. Για τις οικονομικές και εμπορικές σχέσεις εδώ δίνουμε σημασία αξιόπιστες, ε, στο αξιόπιστο επενδυτικό κλίμα. κλίμα που είναι κάτι ιδιαίτερα σημαντικό για τις χώρες της Κεντρικής Ασίας, την καταπολέμηση της διαφθοράς, όπως υπόθηκε και προηγουμένως η διαφθορά είναι πολύ διαδεδομένη και στις πέντε χώρες της Κεντρικής Ασίας και η διασύνδεση με την διεθνή επιχειρησιακή κοινότητα και η περιφερειακή ολοκλήρωση. Τέλος για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Υπήρξαν μεν θετικέ εξελίξει σε ορισμένες χώρες, όπως νομοθετική μεταρρύθμιση και προσπάθειε αποφυγή των βασανισμών, και χρήση τη παιδική εργασία, αλλά η κατάσταση ω προ τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι πολύ ανισχυτική στι περισσότερε χώρε τη Κεντρική Ασία και ενισχύουμε εδώ τι προσπάθειε μα, όπω ξέρετε έχουμε δομημένο διάλογο με, για ανθρώπινα δικαιώματα και με τι πέντε χώρε τη Κεντρική Ασία, ώστε να υπάρχει μια πιο τακτική συνεργασία και ανταλλαγή απόψεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις παραβιάσεις τους και για μεμονωμένες περιπτώσεις. Οι συζητήσεις αυτές είναι πολλές φορές δύσκολες και δεν οδήγησαν κάθε φορά σε ουσιαστικά αποτελέσματα. Παρόλα αυτά είναι πολύτιμες διότι τουλάχιστον επιτρέπουν τη συζήτηση αυτών των ευαίσθητων θεμάτων με δομημένο τρόπο. Τώρα τι κάνει η αντιπροσωπεία μας στην Κεντρική Ασία. Οι αντιπροσωπείες μας έχουν τακτικό διάλογο με αγωνιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και παρακολουθούν τις υποθέσεις δικών και διώξεων και τη δραστηριότητα των ακτιβιστών εκεί και διοργανώνουν σεμινάρια με την κοινωνία των πολιτών. Χωρίς βέβαια να θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή των αγωνιστών. Τέλος υποστηρίζουμε τη δουλειά μη κυβερνητικών οργανώσεων όπως το Ευρωπαϊκό Εργαλείο Δημοκρατίας και σε πλαίσια της ε, πρωτοβουλίας για το κράτος δικαίου στην Κεντρική Ασία οργανώνουμε επαφές και διαλόγους και, με πέντε, και στις πέντε χώρες της Κεντρικής Ασίας με θέματα όπως πρόσβαση στη δικαιοσύνη, ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, ενίσχυση της, των επαγγελμάτων που ασχολούνται με το δικαστικό κλάδο κλπ. Ευχαριστούμε, τελειώνει και αυτό το θέμα. Η διορία κατά διδρομολογιών λίγη στις 23 και η ψηφοφορία θα γίνει στις 10 Δεκεμβρίου. Προβλέπουμε να περάσει την Ολομέλεια τον Μάρτιο. Τώρα το 13 η Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ Ένωσης και της, ε, της ε, Ευρωπαϊκής Οργάνωσης Ατομικής Ενεργείας στο Κοτσιφοπέδιο. Η διαπραγμάτευση άρχισε από τον Οκτώβριο του 2013 μέχρι τον Μάιο. Η συμφωνία υπογράφηκε στις 27 Οκτωβρίου στο Στρασβούργο και το Κοινοβούλιο έλαβε το επίσημο αίτημα από το Χέντε Νοεμβρίου. Η Βουλή του Κοτσιφοπεδίου ενέκρινε επίσης το αίτημα και οι συστάσεις είναι για το τέλος του χρόνου οι επίσημες συστάσεις για την έγκριση από την Ένωση. Το λόγο έχει τώρα ο εισηγητής για το σχέδιο γνωμοδότησής του, ο κ. Σένφιλτ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όντως, όπως είπατε κι εσείς, αυτό, ε, αυτή η συμφωνία σύνδεσης ε, μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ΕΚΑΧ και του Κωσυφοπεδίου ε, 27 Οκτωβρίου μετά από διετής διαπραγματεύσεις. Η συμφωνία αυτή προβλέπει ενισχυμένη συνεργασία και των δύο πλευρών και σε διμερές και σε περιφερειακό επίπεδο και βασικός στόχος είναι η εμβάθυνση των ε, εμπορικών και οικονομικών σχέσεων με το κοσυφοπαίδιο και ένα από τα όργανα ε, για τη διεύρυνση αυτών των σχέσεων είναι η ζώνη ελεύθερων συναλλαγών. Επίσης προβλέπει εναρμόνιση και των, ε, ε της νομοθεσίας του οικοσυφοπεδίου που θα λάβει υπόψη και το κοινωτικό κεκτημένο. Επίσης τονίζει η ανάγκη μεταρρυθμίσεων και η δημιουργία προϋποθέσεων για την προσέλκυση επενδύσεων και τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης. Στο πλαίσιο του, της μεταναστευτικής κρίσης θα πρέπει να γίνει μια συγκράτηση της ε, εξόδου της των μεγάλων μεταναστευτικών ροών από το Κωσυφοπαίδιο προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, το θέμα του καθεστώτος του Κωσυφοπεδίου δεν επηρεάζει τη συμφωνία, ούτε το θέμα της αναγνώρισης από την Ευρωπαϊκή Ένωση της ανεξαρτησίας ε, του κοσυφοπεδίου. Βέβαια, το κοσυφοπέδιο είναι από τις ε, φτωχότερες χώρες της Ευρώπης και ο πληθυσμός των 2 εκατομμυρίων ε, δύσκολα χωρίς βοήθεια θα μπορέσει να δημιουργήσει δημοκρατικούς θεσμούς και να αποκαταστήσει την ευημερία. Και αν δεν το καταφέρει θα αναζητήσει καλύτερη τύχη στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές ε, χώρες. Γι' αυτό και είναι και προς το δικό μας συμφέρον και προς το συμφέρον του Κωσυφοπεδίου να βοηθήσουμε την χώρα αυτή. Σας ευχαριστώ Νίκολα Ιντάντε από το S&D. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή τον κύριο Σέινφελντ για την έκθεσή του και όπως αναφέρεται ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλείται να δώσει την γνωμάτευσή του για την σύναψη συμφωνίας ε, σύνδεσης και εταιρική σχέση με το Κωσυφοπαίδιο για να ξεκινήσει μια νέα φάση στη σχέση με τη χώρα αυτή. Και μάλιστα αυτή η συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεση είναι η τελευταία που έχουμε με χώρα των Δυτικών Βαλκανίων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει στενές ε, οικονομικές σχέσεις με τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και μάλιστα το Μαυροβούνιο και η Σερβία βρίσκονται στον προθάλαμο της ένταξης. Ενώ και οι υπόλοιπες χώρες, ε, Αλβανία, Φιρόμ, θεωρούνται ως ε, δυνητικές υποψήφιες χώρες. Οπότε θέματα ανταγωνιστικότητας, ε, κρατικών προμηθειών, πνευματική ε, ιδιοκτησίας και προστασίας των καταναλωτών είναι πολύ σημαντικά για την εσωτερική μας αγορά και για τις εμπορικές μας σχέσεις με τρίτες χώρες. Και η πολιτική συνεργασία που προβλέπει η Συμφωνία σταθεροποίηση και Σύνδεσης θα πρέπει να εγκαθιδρύσει μία ζώνη ελεύθερων συναλλαγών που θα βοηθήσει την οικονομική ανάπτυξη της χώρας και την αποκατάσταση της σταθερότητας. Θέλουμε εμβάθυνση των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κωσυφοπεδίου υπό την επιφύλαξη βέβαια των εθνικών απόψεων σε ό,τι αφορά το καθεστώς του Κωσυφοπεδίου. Ελπίζω πάντω ότι η γνωμοδότηση θα εγκριθεί με συντριπτική πλειοψηφία. Ευχαριστώ. Ο κύριο Μπούχνερ είναι ο σκιώδη από του πράσινου και έχει το λόγο. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε το λόγο. Άξιο ότι με κύριε εισηγητή. Σα ευχαριστώ πολύ για το σχέδιο και θεωρώ ότι πολλά θετικά στοιχεία περιλαμβάνει. Θα ήθελα να εκφράσω κάποιε αμφιβολίε, ωστόσο. Η μεταβατική φάση 10 ετών για την απελευθέρωση των προϊόντων είναι κάτι πολύ θετικό. Αλλά εγώ προσωπικά θα ήθελα να υπάρχει μεγαλύτερη μεταβατική περίοδος προκειμένου να αποτυπωθεί ακριβώς η πολυπλοκότητα της εφαρμογής ε, των δομών αυτών. Σε ό,τι αφορά τον ε, ε, τομέα των πέντε ετών όπου όλες οι εταιρείες ε, που έχουν έδρα στο Κωσυφοπέδιο θα πρέπει να έχουν τις ίδιες ε, διαδικασίες ε, για δημόσιες συμβάσεις, θεωρώ ότι αυτό καταστρέφει τις δομές και τις εθνικές εταιρείες. Οι ευρωπαϊκές εταιρείε βέβαια μπορεί να κάνουν πιο πολλές δουλειές, αλλά γιατί προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή την προσέγγιση θα βλάψει αυτό την τοπική οικονομία και θα αποδεκατήσει την οικονομία της χώρας και έχουμε μεγάλες αμφιβολίες σε ό,τι αφορά την κατάργηση των ε, ε τελωνιακών δασμών σε ό,τι αφορά τη μείωση των ε, φυσικών ε, πόρων του Βοξίτη πρόκειται για μια, ένα από τους λίγους κλάδους που συντηρούν την οικονομία. Θα ήταν πάρα πολύ επικίνδυνο λοιπόν για το κοσυφοπέδιο να πάυσουν τα έσοδα αυτά και είμαστε κατά των μέτρων αυτών λοιπόν εμφανώς και καταφανώς. Θα θέλαμε λοιπόν να θέσουμε και δύο ερωτήσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε ποιο βαθμό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον τομέα της γεωργίας έχει λάβει υπόψη τις ανησυχίες της χώρας δεδομένης και της σημασίας του κλάδου για την οικονομία της χώρας. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι έχει προσφέρει σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στην αγορά στον κλάδο αυτό και προκειμένου να ε, προστατεύσει τον κλάδο αυτό στο πεδίο. Επίσης θα θέλαμε να μάθουμε κατά πόσον η ρήτρα προστασία στις συμφωνίες με την ε, βιομηχανία ισχύουν και για την γεωργία. Κυρία Ισηγητή, νομίζω ότι θα καταλήξουμε σε ένα καλό αποτέλεσμα για την γνωμοδότηση. Ένα καλό αποτέλεσμα όχι μόνο για μας, αλλά και για το πεδίο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος, και έτσι με αυτή την ε, θετική νότα να ρωτήσω κατά πόσο υπάρχει κάποιος άλλος που θέλει να πάρει το λόγο και αν όχι θα δώσω το λόγο στην κυρία Πρόσφατα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου και ιδιαίτερα τον Άνταμ Σέινφελ, τον εισηγητή, για την ε, θετική γνωμοδότηση Ω προ το θέμα αυτό. Όπω ε, είπατε σωστά, η Συμφωνία Σταθεροποίηση και Σύνδεσης αποτελεί σημαντικό βήμα για την περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης Κωσυφοπεδίου. Και είναι και η πρώτη ε, ενοχική σχέση που έχουμε με το Κωσυφοπέδιο σε Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η τελευταία συμφωνία σταθεροποίηση και σύνδεση με χώρα των Δυτικών Βαλκανίων. Τα πλεονεκτήματα είναι πολλά και διάφορα. Πρόκειται για μια σταδιακή ευθυγράμμιση που θα πρέπει να κάνει το κοσυφοπαίδιο στην ομοθεσία του με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και διατάξεις και θα δοθεί μια νέα ορμή στην ε, κοσοβάρικη οικονομία προκειμένου να προσελκύσει επενδύσεις και να προωθήσει τα τοπικά προϊόντα προβλέπεται αναγνώριση, αμοιβαία αναγνώριση των προσόντων προς όφελος των εργαζομένων και των φοιτητών και προβλέπει πλήρη και άμεση πρόσβαση των κοσοβάρικων προϊόντων στην ευρωπαϊκή αγορά διαφυλάσσοντας πάντως ε, κάποιες διατάξεις για την προστασία της ε, τοπικής παραγωγής και την αύξηση της ανταγωνιστικότητάς της. Η μεταβατική περίοδος έχει δεκαετή διάρκεια και είναι η μεγαλύτερη ε, μεταβατική περίοδος πιο μακροπρόθεσμη που έχουμε προβλέψει για βαλκανική χώρα. Αλλά είναι απαραίτητη μια τέτοια μακρά μεταβατική περίοδος για να μπορέσει η χώρα με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες και να αυξήσει την ανταγωνιστικότητά της. Κάτι τέτοιο βέβαια προϋποθέτει και σημαντική ανάμειξη ε, και δέσμευση και της κυβέρνησης που θα διαδραματίσει αποφασιστικό ρόλο κυρίως ε, την ενίσχυση των εξαγωγικών τομέων, τη δημιουργία ποιοτικών υποδομών, την εξασφάλιση της συμμόρφωσης των προϊόντων με τις προδιαγραφές, ώστε να είναι επιλέξιμα τα προϊόντα για εξαγωγή στην κοινοτική αγορά και να εξασφαλίσει και εύρυθμη λειτουργία των αρμόδιων φορέων, κυρίως της αρχής του ανταγωνισμού. Επιπλέον, πρέπει η κυβέρνηση να στηρίξει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την ανάπτυξη μιας ποιοτικής ε, τοπικής παραγωγής προϊόντων. Σε ό,τι αφορά τα γεωργικά προϊόντα, θα σας δοθούν πιο διεξοδικές πληροφορίες για το πώς βλέπουμε την προστασία των γεωργικών προϊόντων του κοσυφοπεδίου. Αν διαβάσετε προσεκτικά τη συμφωνία, βλέπετε ότι τα πιο ευαίσθητα προϊόντα καλύπτουν, ε, τη χάνουν προστασία. Μερικά μάλιστα ξερούνται κιόλα. από τα θέματα της ειδικής πρόσβασης στην αγορά και για τα πιο ευαίσθητα προϊόντα έχουμε προβλέψει τη μεγαλύτερη, μακρύτερη μεταβατική περίοδο, τη δεκαετή, ώστε να μπορέσουν οι παραγωγοί να προσαρμοστούν στην ανταγωνιστική πίεση και να προσαρμοστούν στις προδιαγραφές και τους κανόνες ανταγωνισμού της ενίας αγοράς. Αυτά. Ευχαριστούμε πολύ. Θέλει ο εισηγητής να πει τίποτα, να προσθέσει. Λίγες παρατηρήσεις μόνο. Ευχαριστώ τους συναδέλφους για τα καλά τους λόγια. Και εγώ είμαι αισιόδοξο ότι θα φέρουμε σε αίσιο πέρα στο έργο μας. Και με βάση τις προηγούμενες εμπειρίες από χώρες που προσπάθησαν να προσαρμοστούν στο κοινοτικό κεκτημένο και να είναι υποψήφιοι να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, η δεκαετής μεταβατική περίοδος είναι μεγάλη και περιμένουμε σημαντικές μεταρρυθμίσεις προς όφελος και της τοπικής κοινωνίας και του κοσοβάρικου έθνους. Ε, συνήθως κρατούν πολύ περισσότερο από μια δεκαετία όλες αυτές οι μεταρρυθμίσεις. Χρειάζονται περισσότερες γενιές. Πάντως είναι σημαντικό να έχουμε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα των απαραίτητων μεταρρυθμίσεων. Είναι ο μοναδικός τρόπος για να επισπευστούν αυτές οι μεταρρυθμίσεις. Τώρα, σε ό,τι αφορά το διεθνή χαρακτήρα που θα πρέπει να, αποκτήσει το εμπόριο και οι επιχειρήσεις, υπάρχουν πολλές πιθανότητες και δυνατότητες εξυγχρονισμού των επιχειρήσεων, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει χωρίς την προσέλκυση αλλοδαπών επενδύσεων και αλλοδαπών επιχειρήσεων. Δεν αρκεί το τοπικό κεφάλαιο για τον εξυγχρονισμό αυτό. Χρειάζεται χρειάζονται και ε, νέες, τεχνο, τεχνολογίες, ε, τεχνογνωσία. Χωρίς επενδύσεις τεχνογνωσία και τεχνολογία δεν νοείται ανάπτυξη. Και η πατρίδα που η Πολωνία πέρασε από τη διαδικασία αυτή. Γιατί με τέτοιες διαδικασίες θα έχουμε τελικά θετικά αποτελέσματα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ να την προσοχή των στο ότι είναι πολύ σύντομο το χρονικό διάστημα για τις ε, 23 ε, Νοεμβρίου στις 12 είναι η προθεσμία, στις 10 Δεκεμβρίου θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή και δεδομένου του καταπήγοντος χαρακτήρα ελπίζουμε να πάμε στην Ολομένη το Γενάρη. Και έτσι λοιπόν ολοκληρώνουμε το σημείο αυτό και να περάσουμε στο 14. Έναρξη διαπραγματεύσεων για συμφωνία ελευθερών συναλλαγών Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ισίας. Και όπω θα θυμάστε, η έναρξη των διαπραγματεύσεων ε, ανακοινώθηκε από την Επιτροπό ε, Μάλμστρον στις 13 Οκτωβρίου στην Τίνιδα και οι δύο διαπραγματευτικές ομάδες συναντήθηκαν και μεταξύ 29 20 και 29 Οκτωβρίου. Δεν είναι η πρώτη φορά λοιπόν που το θέμα αυτό έχει τεθεί και θα συζητήσει το θέμα αυτό και με την πρέσβη τη Τινησία. Δεδομένη τη πολιτική ε, σημασία, αποφασίστηκε ε, να καταρτιστεί ένα ψήφισμα και Μαρία Ντεσσαρνέζ είναι η εισηγητρία, η μόνιμη εισηγητρία για τέτοια θέματα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω και το είπατε κι εσείς ότι το θέμα δεν είναι απλώς θέμα ελευθέρων συναλλαγών, είναι πολιτική συμφωνία, όχι μόνο εμπορική πολιτική. Βλέπουμε πόσο σημαντικό είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνδεθεί με την Τινησία για να τη βοηθήσει να αναπτυχθεί και να διατηρήσει μια πολιτική και δημοκρατική σταθερότητα μακροπρόθεσμα. Η Τινησία νομίζω βρίσκεται σε πολύ σημαντική καμπή της ιστορίας της θυμάστε την Επανάσταση και μετά έγιναν σοβαρές προσπάθειες ε, καθίδρυσης της δημοκρατίας και σταθεροποίησης θυμάστε τις προσπάθειες του κουαρτέτου και του σεπένους του για την Τινησία αλλά ταυτόχρονα γνωρίζουμε ότι το γενικότερο πλαίσιο είναι πολύ δύσκολο για την Τινησία και τους Τινήσιους υπήρξαν οι διπλές επιθέσεις στα Σούσα και τον Μπάρντο υπήρξε η πολύ σημαντική οικονομική κρίση τουριστισμού η σταθερά της απειλής της τρομοκρατίας ανισότητες μεταξύ των περιφερειών που αφορούν ιδιαίτερα τους νέους σε ορισμένες περιοχές της Τινησίας, τους νέους που είναι σε τεράστια πλειοψηφία στην ανεργία. Υπάρχουν τα προβλήματα των συνόρων με την ε, Λιβύη Υπάρχει το θέμα των προσφύγων για το οποίο δεν μιλάμε ποτέ ή όχι αρκετά στην Ένωση. Είναι περίπου 1,8 δις ε, ε, εκατομμύρια στην την Ισία και όλα αυτά δημιουργούν τεράστιες δυσκολίες. Νομίζω λοιπόν ότι είναι πολύ σημαντικό να είναι παρούσα η Ένωση στο ραντεβού αυτό. Η, ανταλα... η συμφωνία αυτή όπως σας το είπα δεν είναι μόνο οικονομική αλλά και πολιτική και θα έπρεπε να συμβάλλει στη σταθεροποίηση της τηνήσίας. Είναι πολύ σημαντικό όλοι μαζί να σκεφτούμε πώς μπορεί να πετύχει η συμφωνία αυτή. Πρέπει να ωφελήσει την Τινησία το σύνολο της οικονομίας της και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το σύνολο των Τινησίων. Γι' αυτό στο ψήφισμα αυτό θέλησα να βάλω ολόκληρο κεφάλαιο για τις συνθήκες επιτυχίας, τους επιτυχίας αυτής της συμφωνίας. Ελπίζω να συμφωνήσουν και οι συνάδελφοι. Πρέπει φυσικά να είναι ασύμετρη η συμφωνία αυτή, δηλαδή να βοηθάει περισσότερο την Τινησία και να μην τονίζει τόσο πολύ μόνο τα δικά μας ζωτικά συμφέροντα. Επίσης προοδευτική, δηλαδή πολύ σημαντικό να δεσμευτούμε, να τους βοηθούμε σε όλη τη διαδικασία και να αφήσουμε, αφήσουμε το χρόνο να προσαρμόσουν ορισμένους τομείς της οικονομίας τους όποτε αυτό απαιτηθεί. Επίσης θα πρέπει να είναι συμφωνία που θα ωφελεί στο σύνολο των τυνησίων, όχι μόνο διαφάνεια δηλαδή, προφανώς χρειάζεται να είναι δημόσιες οι διαπραγματεύσεις, αλλά και μόνιμος διάλογος μεταξύ των συμβαλωμένων. Γι' αυτό προτείνω μεταξύ κοινοβουλευτικών, ευρωβουλευτών και την ισίων βουλευτών καθ' όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων να υπάρχει διάλογος για να εξετάζουμε κατά τις διαπραγματεύσεις από το περιεχόμενό τους και τις θέσεις των διαπραγματευτών βέβαια. Νομίζω ότι πολιτικά αυτό είναι πολύ σημαντικό να μην υπάρχει το αίσθημα ότι άλλοι τα διαπραγματεύονται αυτά, εμπειρογνώμονες δηλαδή, και χωρίς να γνωρίζει την κοινωνία στην Τινησία τι γίνεται και γιατί. Αυτό είναι κλειδί νομίζω για την επιτυχία και τρίτη βασική, τρίτος βασικός όρος να ωφελήσει το σύνολο της οικονομίας η συμφωνία, τον εξυγχρονισμό της για να δημιουργηθούν περισσότερες επενδύσεις σε τομείς κλειδιά για το μέλλον, υψηλή τεχνολογία, τουρισμός, ενέργεια και βιολογική γεωργία, όλοι οι τομείς που αφορούν το μέλλον της Τινησίας. Επιμένω πολύ λοιπόν σε αυτό και νομίζω ότι φτάνουμε σε μια πολύ σημαντική καμπή για την Τινησία ότι η συμφωνία αυτή είναι προς το συμφέρον όλων των Τινησίων αλλά και της Ένωσης γιατί αν υπάρχει μια χώρα από τις επαναστατημένες που πρέπει να στηρίξουμε η Τινησία είναι αυτή για να σταθεροποιήσει τη δημοκρατία της αλλά μας χρειάζεται χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση να βρίσκεται στο πλευρό της για να τη βοηθήσει να προχωρήσει να ανοίξει, να εξυγχρονίσει την οικονομία της και αυτό είναι μια προσπάθεια που δεν πρέπει να τη χάσουμε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και θα δώσω το λόγο τώρα στον κύριο του ΕΛΚ, τον κύριο Σαλατότσιο. Ευχαριστώ. Συμμερίζομαι τις παρατηρήσεις της εισηγήτριας, της κυρίας Τεσσαρνές γιατί σήμερα περισσότερο από ποτέ έχουμε το καθήκον να ενισχύσουμε και να αναβαθμίσουμε τέτοιες συμφωνίες σε μια πολύ λεπτή στιγμή αλλά πολύ επίκαιρη γιατί στη χώρα αυτή έχουμε δημοκρατικούς θεσμούς που μπορούν να ενισχυθούν και να εξασφαλίσουν σε μια επικίνδυνη περιοχή μια σταθερότητα. Γι' αυτό και δεν μπορούμε να παραμελήσουμε αυτήν την ανάγκη υποστήριξης. Σημαντική η συμφωνία και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα πιστεύει ότι είναι πολύ σωστά τα σημεία 19, 20, 21, 22 και 23 για την ανάγκη συνεχούς διαλόγου Επιτροπής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα το σημείο 22 για τον καλύτερο έλεγχο της κατάστασης μέσω της εκπόνησης μελετών επιπτώσεων για να γίνει πιο διεξοδική ανάλυση. θα πρέπει να αποφύγουμε καταστάσεις που αποδυναμώνουν την κατάσταση σε ορισμένε χώρες. Η συζήτηση αυτή φαντάζομαι θα συνεχιστεί και στο μέλλον. Τώρα να πω λίγα λόγια για το ενεργειακό κεφάλαιο της συμφωνίας. Η Επιτροπή μας είπε ότι οι συζητήσεις για το κεφάλαιο αυτό αναβάλλονται για επόμενο γύρο διαπραγματεύσεων. Είναι σημαντικό όμως το θέμα της ε, διασύνδεσης και της ενεργειακής λόγω της υψηλής ζήτησης που υπάρχει αλλά και της ανάγκης της διαφοροποίησης ε, των προμηθευτών για να χρησιμοποιηθούν ε, και να αξιοποιηθούν καλύτερα τα συστήματα διασύνδεσης με τις νότιες χώρες. Πάντως, εν γέννη, η έκθεση είναι πολύ καλή και τη συμφωνούμε και την αποδεχόμαστε. Ο κύριος Μορέλ. Ευχαριστώ. Όπως μας υπενθύμησε η συγγήτρια, η συμφωνία αυτή έχει αναφυσβήτητο πολιτικό και πολιτικό χαρακτήρα και στην ειδική κατάσταση που βρισκόμαστε αποκτά και νέες ε, διαστάσεις και αποχρώσεις. Έχουμε το καθήκον να επιτύχουμε και έχουμε το καθήκον να συνάψουμε μια υποδειγματική συμφωνία με την Τινησία. Αυτό το επιβεβαίωσε και η Επίτροπος Μάλστρομ. Μια υποδειγματική συμφωνία κατά ανάγκη θα είναι και ασύμετρη και προοδευτική. Οι διαπραγματεύσει θα γίνουν φυσικά με τη μέγιστη διαφάνεια και σε στενή συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών της Τινησίας. Θέλουμε παράλληλη ανάπτυξη, κάτι που προϋποθέτει προστασία του γεωργικού και βιομηχανικού τομέα της Τινησίας για όσο χρειαστεί, γιατί δεν είναι, ακόμη, δεν είναι έτοιμοι αυτοί οι δύο για ε, ανταγωνισμό με την Ευρωπαϊκή Ένωση, εξασφάλιση της απαραίτητης τεχνογνωσίας και επίσης να παροτρύνουμε το Συμβούλιο να δημοσιεύσει την διαπραγματευτική εντολή του Δεκεμβρίου του 2011 για να λάβουμε γνώση του περιεχομένου πολύ σημαντική και επίκαιρη αυτή η προσπάθεια και θα πρέπει να είμαστε πολύ απαιτητικοί απέναντι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχουν όμως ε, δυνατότητες ε, βελτίωσης. Μιλούμε για ασύμετρη και προοδευτική εφαρμογή. Σίγουρα χρειάζονται αυτά. Μήπως θα πρέπει να το πούμε ιδιαίτερα και στο κεφάλαιο για το γεωργικό κλάδο, για πλήρω, γιατί το πλήρες άνοιγμα των αγορών με περιορισμό μόνο στα ευαίσθητα προϊόντα δεν αρκεί. Θα έλεγα να είναι σταδιακή και προοδευτική αυτή η προσπάθεια, αυτό το, το ανοίγματο των αγορών. Κάτι άλλο που δεν αναφέρεται παρκώς στο κείμενο. Υπάρχει το ιδιαίτερα λεπτό θέμα για την κοινωνία των πολιτών της Τινησίας, είναι το θέμα του ανοίγματο των αγορών κρατικών προμηθειών. Γι' αυτό δεν λέμε τίποτα στο κείμενο. Και όταν μιλούμε για σύμμετρη εφαρμογή, θα πρέπει να αναφέρουμε με σαφήνεια και το σημείο αυτό των ε, δημοσίων προμηθειών. Επίση, το θέμα των κοινωνικών κανόνων και του σεβασμού των κοινωνικών δικαιωμάτων. Το τόνισε η Επιτροπή Μάνουσα στην Τινησία, αλλά δεν αναφέρεται επαρκώ στο κείμενο. Ένα άλλο θέμα που ενδιαφέρει τα μέλη τη Επιτροπή Διεθνού Εμπορίου. Ε, ίσως το διάβασα προσεκτικά το ειδικό κεφάλαιο για την προστασία των επενδύσεων, αλλά νομίζω ότι δεν αναφέρεται αρκετά αυτό το θέμα. Ακόμη και αν καταλήξουμε σε, μια ρήτρα επίκληση διαφορών κράτους επενδυτή στο σχετικό κεφάλαιο για τις επενδύσεις. Πάντως το κείμενο είναι καλό στο μέτρο που λαμβάνει υπόψη το συμβολικό πολιτικό χαρακτήρα που έχει σύναψη μια τέτοια συμφωνίας. Μόνο τον κύριο Φεράν βλέπω από τους υπόλοιπους και ηγητές από το ΙΕΝΕΦ. E Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Από το 2010 και την ανατροπή του προηγούμενου καθεστώτος η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να στηρίξει μια Τινησία που είναι σχεδόν ετοιμοθάνατη που ψυχοραγεί μάλλον και το να το επιχειρούμε με τις εμπορικές μας συμφωνίες δεν νομίζω ότι είναι κατάλληλο γιατί η αποσταθεροποίηση της Τινησίας οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις δράσεις της Γαλλίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και σήμερα για μια ακόμη φορά η γεωργία χρησιμοποιείται ως ε, διαπραγματευτικό εργαλείο μιας ε, πολιτικά αντικής πολιτικής και πάνω από ένα δισεκατομμύρια χρησιμοποιήθηκαν ε, για, του, για τους Γάλλους γεωργούς που θα πρέπει να καλύψουν τα σπασμένα της Τινησίας. 35.000 τόνους ελαιόλαδο θα είναι η αύξηση της ε, αντίστοιχης ποσόστοσης της θυμησίας, ε, κάτι που θα επηρεάσει αρνητικά τις χώρες του Νότου. Και μάλιστα εκπλήσαμε που οι Ιταλοί θέλουν να θεωρήσουν υποδειγματική αυτή τη συμφωνία με την Ισία. Δεν νομίζω ότι οι Ιταλοί παραγωγοί ελαιολάδου θα εκτιμήσουν ιδιαίτερα την αύξηση της ποσότητας ελαιολάδου της Τινησίας. Πάντως η συμφωνία αυτή δείχνει την βούληση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω των συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών να επιβάλλει μια πολιτική ανθρωπίνων δικαιωμάτων που δυστυχώς για μία ακόμη φορά θυσιάζει στο βωμό της ένα ολόκληρο κλάδο της Ευρωπαϊκής Γεωργίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Κυρία Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ μιλώ εξ ονόματος του Πατρίκ Λαγκερίκ που αποσιάζει σήμερα λόγω των γεγονότων του Παρισιού. Λοιπόν, έχει τις εξής παρατηρήσεις. Ως ομάδα είμαστε υπέρ της θέσης της έκθεσης που θυμίζει τη σημασία της Τινησίας για τις σχέσεις μας με τον Μαγράμ και τη σημασία του να βοηθήσουμε την κοινωνία της Τινησίας να ξεπεράσει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει για τον εκδημοκρατισμό της. Είναι σημαντικό να διατηρηθεί η ασύμετρη διάσταση στη συμφωνία αυτή. Για μας είναι σημαντικό. Και η ασυμμετρία αυτή πρέπει να σημαίνει ότι θα αναγνωριστεί το δικαίωμα της Τινησίας να παράγει φαρμακευτικά προϊόντα τοπικά να διατηρήσει τις δημόσιες τις υπηρεσίες έναντι του ευρωπαϊκού ανταγωνισμού και επίσης το δικαίωμά της να νομοθετεί. Οι μηχανισμοί του ESDS λοιπόν και της επίλυσης των διαφορών μεταξύ των διαφόρων επενδυτών και του κράτους πρέπει να βελτιωθούν. Πρέπει να βοηθήσουμε την κοινωνία των πολιτών και ιδιαίτερα τα συνδικάτα τα οποία θα έπρεπε ήδη να έχουν συμμετάσχει περισσότερο στις διαδικασίες στις διαπραγματευτικές διαδικασίες. Αυτό είναι μια έλλειψη λοιπόν που παρατηρούμε. Είναι σημαντικό να γίνει μια παύση μέχρι η κοινωνία των πολιτών της Τινησίας να μπορέσει να συμμετάσχει στη διαδικασία με παράλληλη βέβαια οικονομική, αξιο... κοινωνική και περιβαλλοντολογική αξιολόγηση όλων αυτών. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα το λόγο έχει πάλι η κυρία Ρένα. Euh, euh, ευχαριστώ. Συμφωνώ απόλυτα με τον Εμμανιέλ Μορέλ. Θα ήθελα στο ψήφισμα να συμπεριλάβουμε και την ανάγκη εκπόνησης ε, μελετών επιπτώσεων από την Τινησία με κοινοτική χρηματοδότηση. Αυτό θα ήταν σημαντική τεχνική υποστήριξη προς την Τινησία με συμμετοχή των συνδικάτων και της κοινωνίας των πολιτών. Οπότε είναι σημαντικό τέτοιες μελέτες επιπτώσεων που θα γίνουν από την Τινησία να χρηματοδοτηθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σα Σας ευχαριστώ. Και τώρα θα δώσω το λόγο στην κύριο Πυρογιάννα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να κλείσουμε τη συζήτηση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και πολύ με τιμα το γεγονό ότι μου δίνετε το λόγο όπω και στα μέλη τη Επιτροπή για να σχολιάσω τουλάχιστον τη συζήτηση και τα όσα ακούσαμε έω τώρα. Καταρχά, προφανώ όπω είπατε και εισαγωγικά, αυτή η διαπραγμάτευση μόλι ξεκίνησε τον περασμένο μήνα. Στην την για να διευρύνει ένα ήδη φυστάμενο τομέα ελευθέρου ε, εμπορίου που δημιουργήθηκε στη δεκαετία του 90 μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ισίας που ήδη περιλαμβάνει μια ασυμμετρία σε ό,τι αφορά το εμπόριο και την γεωργία και ήδη προβλέπει αμφίδρομη απελευθέρωση του εμπορίου και των βιομηχανικών προϊόντων μέσω της κατάργησης των ε, δασμών αυτό που θέλαμε να κάνουμε στην Σφαιρική και σε βάθος Συμφωνία Ελευθερών των Αλλαγών με την Τινησία είναι να διευρύνουμε και να εμβαθύνουμε τις σχέσεις μας και με τον τρόπο αυτό να μπορέσουμε σταδιακά να εντάξουμε την ε, ε, οικονομία της Τινησίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην ενιαία αγορά με πλέον εκτήματα και σε ό,τι αφορά την καλύτερη οικονομική διακυβέρνηση αλλά και σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στην αγορά σε θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην Ιστορική και Συμβάθο Συμφωνία Ελευθερών Συναλλαγών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντιλαμβάνεται ασφαλώ όλε ε, τι ανησυχίε και τα ιδιαίτερα ζητήματα που υπάρχουν στην Τινησία σε ό,τι αφορά τη γεωργία και τι υπηρεσίε κυρίω και στη διαδικασία διαπραγμάτευση. Ε, σκοπεύουμε να τα λάβουμε αυτά υπόψη με τον ανάλογο τρόπο. Και όπω πολύ προτείνεται, σκοπός μας θα είναι να προχωρήσουμε με μια προσέγγιση ασύμετρη και βαθμιαία σε ό,τι αφορά και τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων. Και σε συνάρτηση με αυτό θα πρέπει να διευκρινίσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ελπίζει να κινητοποιήσει και τα αντίστοιχα μέτρα, συνοδευτικά μέτρα για να βοηθήσει την Τινησία και κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων και κατά την ε, φάση εφαρμογής στη συνέχεια τη Φερική και Ζεβαστος Συμφωνία Ελευθερών Συναλλαγών. Ελπίζουμε να υπάρχουν και παράλληλε δράσει από τα μεμονωμένα κράτη-μέλη, να μην είναι μόνο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη δικασία αυτή, καθώ και να υπάρξουν ε, δράσει και από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, την ΕΤΕΠ και την Τράπεζα ε, Ανεκοδόμηση. Και προφανώ βρισκόμαστε σε μια διαδικασία η οποία θα πάρει μήνε σε ό,τι αφορά τη διαφάνεια και την ε, συμπερίληψη όλων των φορέων, ένα θέμα που έθιξαν διάφορα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Επιτροπής ε, του Κοινοβουλίου. Από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, θέλουμε ναι, να διασφαλίσουμε καλή ποιότητα και απόλυτη διαφάνεια στη διαδικασία και συνεχή διάλογο με την κοινωνία των πολιτών και στην Ευρώπη αλλά και στην Τινησία. Στις συναντήσεις που έλαβαν χώρα τον περασμένο μήνα και κατά την επίσκεψη της Επιτρόπου Μάλμστροπ και την επόμενη εβδομάδα κατά την εκείνη των διαπραγματεύσεων. Συμμετείχε η κοινωνία των πολιτών στην την και αυτό αναμένουμε ότι θα συνεχιστεί καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας και προφανώς θα συνεργαστούμε ε, στο πλάι των αρχών της γιατί προφανώ κάποιε από τι διαδικασίε διαφάνεια ιδιαίτερα στην Τινησία, θα πρέπει να οργανωθούν από αμφότερε τι πλευρέ. Εντό παρενθέσεων να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με χαρά θα υποστηρίξει και τον διακοινοβουλευτικό διάλογο εφόσον το επιθυμείτε που θα εγκαθιδρυθεί με τι ε, αρχέ τη Τινησίας. Ένα σύντομο σχόλιο τώρα. Επιτρέψτε μου για δύο άλλα σημεία, τα οποία αναφέρθηκαν εν παρόδο. Ναι, αναμένουμε ότι θα υπάρξει κεφάλαιο για την ενέργεια, που θα αποτελέσει ε, τμήμα της σφαιρικής και σε βάθος συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών και αναμένουμε και ένα κεφάλαιο για τις δημόσιες συμβάσεις και για τις ε, επενδύσεις και για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Και δεδομένου ότι βρισκόμαστε σε φάση εισαγωγική των ε, διαπραγματεύσεων, βρισκόμαστε στη φάση παρουσίασης των προθέσεών μας και των ε, προπαρασκευαστικών δράσεων που έχουν λάβει χώρα τα περασμένα χρόνια και αυτό ασφαλώς σημαίνει ότι οι διαπραγματεύσεις θα πρέπει να εξελιχθούν με την ώρα τους. Και σκοπεύουμε να κρατάμε ενήμερη την Επιτροπή σας κατά τη διάρκεια των εξελίξεων. Αυτά, Πρόεδρε, και προφανώ θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε τη συζήτηση με μεγάλο ενδιαφέρον και να ανταλλάσσουμε απόψει. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρο, και ασφαλώ σα θεωρούμε εισάξιου να δώσω το λόγο στην κυρία Μαρία Ελδεσόνης για να απαντήσει. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συμφωνώ σχεδόν με το σύνολο, όχι όλους βέβαια, αλλά με τους περισσότερους από όσους μίλησαν. Οι συνάδελφοι του ΕΛΚ έφυγαν τώρα. Συμφωνώ ότι παρά το ότι το κείμενο λέει μερικά πράγματα θα μπορούσαμε να τα ενισχύσουμε. Η ιδέα ας πούμε χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση συμφωνώ απόλυτα. Ο μόνιμος διάλογος που αναφέρθηκε επίσης συμφωνώ της διασύνδεσης για τα ενεργειακά είναι κάτι που επίσης δεχόμαστε. Με τον Εμμανουέλ Μορέλ τα ίδια συμφωνούμε απόλυτα. Φυσικά ζητούμε τη δημοσίευση της διαπραγματευτικής εντολής. Καιρός θα ήταν το Συμβούλιο να τα καταλάβει αυτά κάποτε. Τον κοινωνικό διάλογο μπορούμε να τον ενδυναμώσουμε, την προστασία των επενδύσεων επίσης συμφωνώ και θα δούμε τι τροπολογίες θα μπορούσαμε να καταθέσουμε σχετικώς όπως και για την προστασία ορισμένων συγκεκριμένων τομέων και το προοδευτικό άνοιγμα για τα γεωργικά προϊόντα. Επίσης συμφωνώ με τη διατήρηση των δημοσίων υπηρεσιών και τη σύνδεση την καλύτερη δυνατή με την κοινωνία των πολιτών στην Ισία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι μάλιστα κλειδί για την επιτυχία της συμφωνίας. Άλλος συνάδελφος μίλησε για το κόστος που θα έχουν όλα αυτά που πρέπει να είναι σοβαρή όσο για το ελαιόλαδο 70.000 το πολύ εξάγει την Ισία ενώ πάνω από 1,5 εκατομμύριο η Γαλλία. Το την Ισιακό ελαιόλαδο είναι πολύ καλής ποιότητος, σας συνιστώ να το δοκιμάσετε είναι ελαιόλαδο που το εκτιμούν ιδιαίτερα και οι αγορές και η Ιταλία που χρησιμοποιείται πολλές φορές για να βελτιώσει την ποιότητα του Ιταλικού ελαιολάδου. Σε όλους συμφέρει δηλαδή. Πάντως, στην εποχή μας δεν είναι σωστό να στρέφουμε τους λαούς τον ένα κατά του άλλου. Δεν είναι η καταλληλότερη μέθοδος. Αυτά κύριε Πρόεδρε και σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Ολοκληρώνουμε τη συζήτηση. Χρονοδιάγραμμα. 15 Δεκεμβρίου στις 12 λίγη προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών. 25 Ιανουαρίου θα γίνει ψηφοφορία στην Επιτροπή και κάποια στιγμή αργότερα στην Ολομέλεια. Περνάμε στο σημείο 15, ανταλλαγή απόψεων για την αναδιατύπωση του κανονισμού πρόσβασης, ε, ελεύθερης πρόσβασης στην αγορά. Πρόκειται για προϊόντα χωρών και που προβλέπονται συμφωνίε οικονομική εταιρική σχέση ή συμφωνίε που οδηγούν στη σύναψη τέτοιων συμφωνιών. Πρόκειται για αναδιατύπωση. Η συγκεκριτή μα είναι ο κύριο Βαγουένσα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τι έχουμε εδώ. Έχουμε μια κωδικοποίηση και αναδιατύπωση του κανονισμού του Συμβουλίου, του λεγόμενου κανονισμού για την πρόσβαση στι αγορέ. Πρόκειται για το νομικό μέσο που προβλέπει ε, την ε, αντιμετώπιση κάποιων εμπορικών προβλημάτων ε, για σύναψη ή προετοιμασία σύναψη συμφωνιών οικονομικής συνεργασίας και προβλέπει αδοσμολόγητη και άνευ ε, ποσοστό σε πρόσβαση στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μεταβατική περίοδο που χρειάζεται για την υπογραφή και κύρωση τέτοιων συμφωνιών οικονομικής εταιρικής σχέσης. Ε, το 2007 εγκρίθηκε ο κανονισμός ε, ο αρχικός. Έχει τροποποιηθεί πολλές φορές και τώρα μετά την ευθυγράμμιση με τη συνθήκη της Λισαβόνας για το Γενικό Νόμο για το Εμπόριο και τις επακόλουθες εξουσιοδότηση για τους επακόλουθους κατοξιδότηση κανονισμούς ε, προβλέπεται ευθυγράμμιση με το κοινοτικό κεκτημένο και με την τελευταία κωδικοποίηση εξασφαλίζεται σαφήνεια και ευανάγνωστο του κανονισμού με απλούστευση της κοινοτικής νομοθεσίας. Ταυτόχρονα χρησιμοποιούμε τη μέθοδο της αναδιατύπωσης προκειμένου να τροποποιήσουμε το κείμενο σε, μερικές, ε, σε μερικά σημεία. Η πιο σημαντική αλλαγή προτείνει την, την αλλαγή στην κατεξοδότηση πράξης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να μπορεί να υιοθετεί τις πράξεις που θα εφαρμόζονται σε προϊόντα προέλευσης Νοτιού Αφρικής. Χρειάζεται αυτό μέχρι όταν εγκατασταθούν οι σχετικές δια... διατάξεις για το εμπόριο, την ανάπτυξη και τη συνεργασία. Και ε, τις σχετικές διατάξεις Συμφωνίας Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και μερικών ε, χωρών της Μεσηβερινής Αφρικής που συνήθει στις 15 Ιουλίου του 2014. Το κείμενο είναι έτοιμο για υπογραφή και κύρωση. Δεύτερη αλλαγή σημαντική αφορά το άρθρο 22. Εκεί γίνεται μνήμα του άρθρου 134 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας η διαγραφή αυτή θα πρέπει, η αναφορά συγγνώμη αυτή θα πρέπει να διαγραφεί, γιατί το ίδιο το άρθρο 134 καταργήθηκε με τη θέση σε ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας. Και η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων έχει εκδώσει ευνοϊκή γνώμη και επιβεβαιώνει ότι η πρόταση είναι απλή κωδικοποίηση και περιορίζεται σε συγκεκριμένε ε, ουσιαστικές τροποποίησεις. Γι' αυτό και προτείνω ως εισηγητής να εγκρίνουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής χωρίς περαιτέρω τροποποίησης. Ευχαριστώ. Θέλει άλλος κανείς το λόγο? Ποιος έχει μείνει? Ναι, ναι. Συμφωνώ πάντως με την τελευταία σας σύσταση να εγκρίνουμε την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής χωρίς τροποποίησης. Και να δώσω το λόγο στην κυρία Στέμα την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το σημείο αυτό. Τον κύριο μάλλον, συγγνώμη. Αν θέλει να πει κάτι. Ή δεν υπάρχει καν εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το σημείο αυτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η Επιτροπή συμμερίζεται την άποψη κ. Βαλέντσα, ότι πρέπει να προχωρήσουμε γρήγορα και χωρίς πρόβλημα. Πολύ ωραίος συνενετικός τρόπος να τελειώσει η συνεδρίασή μας. Τελειώνει αυτό το θέμα λοιπόν. Η διορία κατάθεση τροπολογιών είναι 24 Νοεμβρίου στις 12 το μεσημέρι. Ευχαριστούμε τον εισηγητή. Το 16 έχει αναβληθεί. Τώρα τα διάφορα δεν έχει. Επόμενη συνεδρίαση 30 Νοεμβρίου στις 3 και 1η Δεκεμβρίου στις 9 στις 15 η ώρα σας. Κατευχαριστώ για την προσοχή.